Κυρίες και κύριοι, Σας παρακαλώ λίγη ησυχία. Συνεχίζουμε τις εργασίες της Επιτροπής Προπολογισμών. Έχουμε μία ώρα για την παρουσίαση της κατάστασης των αποκεντρωμένων οργανισμών και το πρόβλημα της χρηματοδότησης των δραστηριοτήτων τους την επόμενη χρονιά, μέσα στο 2013. Κάθε χρόνο γίνεται αυτή η συνάντηση. Έχουμε ανταλλαγή απόψεων εδώ στην Επιτροπή Προϋπολογισμών, όπου η Τρόικα των Διευθυντών Δηλαδή, τρει διευθυντέ που εκπροσωπούν το σύνολο των οργανισμών έρχονται εδώ και συζητούν μαζί μα. Στο φάκελό σα έχετε όλα τα έγγραφα που υπάρχουν. για να γίνει αυτή η συζήτηση. Και για να εκτιμήσετε τα όσα θα ακούσετε. Επίσης, λάβαμε υπόψη μας την ψηφοφορία που έγινε στο Κορεπέρ για το σχέδιο προπολογισμού του 2013. η ψηφοφορία αυτή, το αποτέλεσμα της ψηφοφορίας θα πάει στο Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών και κατά 99,999% οι Υπουργοί επιβεβαιώνουν τον τρόπο που ψήφισαν στο Κορεπέρ οι εκπρόσωποι. Η ψηφοφορία αυτή είναι πολύ αυστηρή σε ό,τι αφορά τον προπολογισμό των οργανισμών. Γίνεται μια μικρή διαφοροποίηση ανάμεσα στις υπηρεσίες που φτάσαν στην ταχύτητα πλεύσης και στις υπόλοιπες ε, υπηρεσίες και οργανισμούς. Λαμβάνοντας υπόψη, οι παλιοί οργανισμοί έχουν λάβει νέα καθήκοντα. Και λαμβάνοντας υπόψη επίσης, το γεγονός ότι κάποιοι οργανισμοί είναι εντελώ καινούργοι και επομένως θα χρηματοδοτηθούν για πρώτη φορά. Συνολικά πάντως το γενικό κλίμα δεν χαρακτηρίζεται από δημοσιονομική γενεοδορία για τις δαπάνες, τις λεγόμενες, της κατηγορίας ε, Και φυσικά τα περισσότερα κονδύλια των οργανισμών αφορούν αυτή την κατηγορία. Καλώς ορίζω τον κύριο Γκέρτς από την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία, μάλλον τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Χημικών Ουσιών που βρίσκεται εδώ στην πρώτη σειρά, στο πρώτο έδρανο. Το χαιρετίζουμε, τον κύριο Μίκαλε Χέμπορκ από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Σιδηροδρόμων, καλώ ήρθατε, και ο κ. Ντάνκαν από το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την πρόληψη των ασθενειών και τον έλεγχο των ασθενειών. Αυτή είναι η Τρόικα, λοιπόν, με τη μεσογειακή έννοια του όρου, δηλαδή γενναιόδορη. Η κυρία Κρίστα Ζετλάτσεκ, που είναι Διευθύντρια της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας για την ασφάλεια και την υγεία στο χώρο εργασία, Πού είναι η κυρία αυτή. Α, γεια σας. Καλησπέρα. Ο κ. Πάτρι Γκούντου. Μου στείλε... Μου ζητάει συγγνώμη, δεν είναι παρόν, ένα συνεργάτης του θα τον εκπροσωπήσει. Και καλωσορίζω επίσης και τα άτομα που ανήκουν σε άλλες υπηρεσίες, σε άλλους οργανισμούς και που θα συνεισφέρουν στη συζήτηση. Ξέρουμε μια δημόσια συνεδρίαση αυτή εδώ. Φυσικά αυτή η συζήτηση θα ολοκληρωθεί με την παρουσίαση της Utah Hawk, που είναι η δική μας εισηγήτρια. Η ειδική εισηγήτρια. Και τον εισηγητή για τον προπολογισμό του 2013, που είναι ο Τζοβάνι Λαβία. Η βασική παρουσίαση θα γίνει από τον κύριο Ντάνσετ. Του δίνω το λόγο λοιπόν και ζητώ από όλου τους ομιλητέ να είναι σύντομοι και λακωνικοί. Γιατί 16, 16 ακριβώς, δηλαδή 4 ώρα το απόγευμα, πρέπει να σταματήσουμε αυτή τη συζήτηση. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητά μέλη τη επιτροπή. Χαίρομαι που έχουν ευκαιρία να ανταλλάξουμε σας απόψη για τον προπολογισμό του 2013. Ζητήσατε από τι αποκεντρωμένε υπηρεσίε να δώσουν συγκεκριμένα παραδείγματα για τον αντίκτυπο που θα έχει το σχέδιο προπολογισμού τη Κομισιόν για το επόμενο έτο. Στο έγγραφο που σα στείλαμε πριν από την συνεδρίαση δίνουμε τέτοια παραδείγματα. Πρέπει όμω να τονίσω πω αυτά τα παραδείγματα δεν ε, ε, λαμβάνουν πλήρω υπόψη τι πρόσφατε θέσει του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Όπω ξέρετε, το Συμβούλιο ζητά περαιτέρω μειώσει του προσωπικού και τη επιδότηση, ειδικά για τι νέε υπηρεσίε και αυτέ με τα νέα καθήκοντα. Για να φέρω κάποια παραδείγματα. Μείον 10 θέσει στην υπηρεσία αξιογράφων, μείον 6 από την Ευρωπαϊκή Τραπεζική Αρχή, μείον 10 από την υπηρεσία φαρμάκων, ασφάλεια ασφάλεια μείον 32 υπηρεσία περιβάλλοντος μειών 3 και η νεότερη υπηρεσία για την διαχείριση πληροφοριακών συστημάτων δικαιοσύνης και στον τομέα της δικαιοσύνης και εσωτερικών επίσης αρκετέ μειώσει. Μείον 11. Επίση, μιλάμε για μειώσει των προπολογισμού στου τίτλου 1 και 2, κατά το οποίο βεβαίω ανατρέπει την ισορροπία, γιατί έτσι δεν υπάρχει δυνατότητα να διαθέσουν επιχειρησιακά κονδύλια στον τίτλο 3 και αυξάνεται η ανάγκη για τις ε, μεταφορές κοντιλίων που ζητάμε. Επίσης, πολλές υπηρεσίες θα έχουν νέα καθήκοντα το 2013. Ήδη υπήρχε πρόβλημα από αυτά τα οποία πρότεινε η Κομισιόν και οι δε περικοπές του Συμβουλίου δημιουργούν δυσκολίες για την εκπλήρωση των εντολών αυτών. Αυτά αφορούν την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία για την Ασφάλεια της Αεροπορίας, το Ευρωπαϊκό Ίδρυμα Περιβάλλοντος εκπαίδευση Φαρμάκων, τη Frontex, τη Europol και την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Χημικών Ουσιών τη οποία είμαι εκτελεστικό διευθυντή. Είμαστε σε ιδιαίτερη θέση καθώ ο νέο κανονισμό για τα βιοκτώνα, το οποίο υιοθετήθηκε, μα απαγορεύει να χρησιμοποιήσουμε άλλη γραμμή του προπολογισμού για τι αστηριότητε βιοκτώνων. Οπότε, αν γίνονται εκτές οι που προτείνονται από το Συμβούλιο, δεν μπορώ να εγγυηθώ την σωστή ε, λειτουργία του κανονισμού αυτού. Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων ε, Ασφαλείας ε, της Αεροπορίας, η Frontex και η Υπηρεσία Ασύλου έλαβαν ακόμη λιγότερους πόρους από αυτού ε, οι οποίοι απαιτούνται για τη σωστή λειτουργία. Παραδείγματο χάρη, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Φαρμάκων πρέπει να εφαρμόσει τη νέα νομοθεσία φαρμακοϊπαγρύπνηση από τον Ιούλιο. Κάτι το οποίο δεν θα μπορέσει να κάνει με τι περικοπέ προσωπικού όπω προτείνονται για το 2013. Συμπερασματικά, εάν περάσει η θέση του Συμβουλίου και γίνουν ακόμα μεγαλύτερε περικοπέ, πολλέ υπηρεσίε δεν θα μπορέσουν να κληρώσουν την εντολή την οποία έχετε δώσει εσείς ως Ευρωπαίος νομοθέτης. Είναι σωστό οι εκτελεστικοί διευθυντές ε, να πρέπει να αποφασίζουν ποια τμήματα της εντολής δεν μπορούν να εκπληρώσουν. Εμείς έχουμε πραγματικά το δικαίωμα να αγνοήσουμε καθήκοντα τα οποία μας ανέθεσε ο νομοθέτης. Πρέπει να πω πως εγώ και οι συναδελφοί μου δεν ε, νιώθουμε πάρα πολύ καλά με κάτι τέτοιο. Κομισιόν και Συμβούλιο βλέπουν ε, τους πόρους για όλες τις υπηρεσίες ως έναν ενιαίο φάκελο δημοσιονομικό. Αυτό το οποίο σημαίνει πως όταν δημιουργείται μια τέτοια υπηρεσία αυτομάτως κόβονται πόροι από τις άλλες. Αλλά τα καθήκοντα παραμένουν τα ίδια. Οι υπηρεσίες δεν είναι νομοθετικά θεσμικά όργανα τα οποία μπορούν να λάβουν απλά λιγότερες ε, πρωτοβουλίες. Έχουμε εντολές οι οποίες επηρεάζουν άμεσα εταιρείες και πολίτες. Και η μεγαλύτερη ανησυχία μας είναι το πολιετές μεσονομικό πλαίσιο της Ένωσης. Εάν οι υπηρεσίες αυτές συνεχίζουν να αντιμετωπίζοντας ένας ενιαίος μεσονομικός ε, φάκελος, ανησυχούμε για το αποτέλεσμα. Αυτό το οποίο φοβόμαστε είναι πως κάποια στιγμή σε κάποιο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα κλείσει μια συμφωνία αργά τη νύχτα ε, που θα έχει τεράστιες αυθαίρετες περικοπές χωρίς να δοθεί καθόλου σκέψη στο πώς πρέπει να εφαρμοστούν αυτές οι περικοπές. Οι υπηρεσίε και τα ΔΕΛΤΑ κατόπιν θα πρέπει να, κάνουν, να λάβουν σημαντικές αποφάσεις χωρίς καμία κατεύθυνση από αυτούς οι οποίοι λαμβάνουν τις αποφάσεις. Ζητώ λοιπόν από την Επιτροπή Προπολογισμού να μην επιτρέψουν να συμβεί κάτι τέτοιο. Αρχίζοντας από φέτο, θα μπορέσετε να δώσετε μια πιο έξυπνη προσέγγιση των προπολογισμών αυτών. Και στόχος θα πρέπει να είναι το τι περιμένουν από μας οι πολίτες και το πώς θα πρέπει να συνεργαζόμαστε με τους ε, εταίρους μας. Γιατί σε πολλέ περιπτώσει μειώνεται το συνολικό κόστος για το φορολογούμενο τη υπηρεσία μας. Συχνά είναι φθηνότερο να γίνει κάτι μία φορά στο ευρωπαϊκό επίπεδο, αντί να γίνει 27 φορές σε εθνικό επίπεδο. Συμπερασματικά, σκοπεύουμε λοιπόν και αυτό το οποίο ζητάμε είναι να εξετάσετε κατά περίπτωση τις ε, υπηρεσίε αυτέ. Ξέρω πω το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σκοπεύει να έχει ένα προπολογισμό ανάλογο των φιλοδοξιών τη Ευρωπαϊκή Ένωση και σα στηρίζουμε. Είμαστε σύμμαχοί σα όταν ζητάτε έναν κατάλληλο και επαρκή προπολογισμό. Το δίκτυο των υπηρεσιών που είναι εδώ πέρα παρόν είναι στην διάθεσή σα για να διευκολύνει αυτόν τον σημαντικό διάλογο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πολύ ωραία. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Τα άλλα μέλη της Τρόικα θα ήθελαν να πούν κάτι. Όχι. Σας ευχαριστώ. Πολύ σαφής παρουσίαση, ολοκληρωμένη, λιτή. Υπάρχουν ερωτήσεις ή σχόλια. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα ήθελε να αιτιολογήσει τις προτάσεις και να σχολιάσει την ψήφο του Κορεπέρ, ο κύριος Πρέσα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να εξηγήσω κάπως την πρόταση της Κομισιόν και να σας δώσω μερικά συγκυριακά στοιχεία που θα μπορούσαν να πλαισιώσουν τη συζήτηση. Αριθμοί οι αποκεντρωμένοι οργανισμοί αποτελούν ένα δυναμικό τμήμα στην στο, στο σχήμα μάλλον των ευρωπαϊκών οργάνων και οργανισμών και για το 2013 έχουμε 5.115 θέσεις εδώ δεν εντάσσονται τα, οι 820 θέσεις των αυτοχρηματοδοτούμενων οργανισμών, φτάνουμε δηλαδή πάνω κάτω στις 6.000 θέσεις, 1.500 αποσπασμένους ε, υπαλλήλους ή συμβασιούχους έχουμε επίσης Περίπου δηλαδή συνολικά είναι 7.500 κεφάλια για το 2013. Τώρα η Κομισιόν ε, επέβαλε διακρίσεις στους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Όχι, δεν αντιμετώπισε τους, όλους τους οργανισμούς κατά τον ίδιο τρόπο. Όπως θα θυμάστε, η Κομισιόν έδωσε έναν προσανατολισμό και για τα θεσμικά όργανα και για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς για προσπάθειες αποτελεσματικότητας και μείωση κατά 1% του προσωπικού των θεσμικών οργάνων. Το εφάρμοσε και στην ίδια την Κομισιόν αυτό. Το αποτέλεσμα για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς είναι 257 θέσεις παραπάνω. Και αυτό το αντισταθμίσαμε με μία μικρή μείωση σε οργανισμούς οι οποίοι ήδη λειτουργούν εύρυθμα, βρίσκονται εμπλό, υπέρ των νεοσύστατων οργανισμών και των οργανισμών εκείνων που ανέλαβαν νέες αρμοδιότητες για το θέμα της ταξινόμησης. Ποιο είναι το κριτήριο το οποίο χρησιμοποιεί η Κομισιόν για να ταξινομήσει τους οργανισμούς, δηλαδή ήδη λειτουργούντες οργανισμοί έμπλο, ε, νέοι οργανισμοί και νέες αρμοδιότητες. Το κριτήριο είναι ότι η ανάθεση νέων αρμοδιοτήτων σημαίνει ένα νέο κονδύλι με ανακοίνωση της Επιτροπής. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε μία επίσημη πρόταση που υποβάλλεται στο Συμβούλιο και στο Κοινοβούλιο και εξετάζεται βάσει του άρθρου 47 της Διαθεσμικής Συμφωνίας. Έχουμε λοιπόν μία επίσημη φάση, ένα επίσημο στάδιο ε, για τη δημιουργία νέων οργανισμών ή για οργανισμούς που αναλαμβάνουν νέες αρμοδιότητες ε, που μας επιτρέπει να δούμε αν είναι σύμβατα όλα αυτά με την οροφή των δαπανών στην ε, κατηγορία στην οποία εντάσσονται. Τώρα, για τον προϋπολογισμό για τους αποκεντρωμένους οργανισμούς. Γιατί εμείς λαμβάνουμε υπόψη μας αυτόν τον νέο παράγοντα. Εμείς εγγράφουμε στον προϋπολογισμό πιστώσεις αλλά όχι με σκοπό να δημιουργήσουμε αποθέματα τα οποία δεν θα χρησιμοποιούνται. Το πλεόνασμα των οργανισμών καταγράφεται ως διαθέσιμο εισόδημα για την επόμενη χρονιά. Οπότε το νοπό χρήμα το οποίο έρχεται από τον προϋπολογισμό μας επιτρέπει να εξισορροπούμε τα έξοδα με, τις, ε, τα έσοδα. Εμείς, ε, εγώ άκουσα να μιλάμε πολύ εδώ για μείωση θέσεων. Δεν είναι μείωση, είναι απλώς λιγότερη αύξηση. Έχουμε 257 υπαλλήλους πλέον στο σχέδιο προϋπολογισμού. 2013. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Γιούτα θέλετε το λόγο τώρα. Μετά, οκ. Okay. Ιαν. Ευχαριστώ για την παρουσίαση από τον Διευθυντή του Οργανισμού, τον εκπρόσωπο της Τρόικα και από την Κομισιόν. Είπατε ότι οι οργανισμοί μπαίνουν σε μία κατηγορία, αλλά θεωρούμε όλες αυτές τις δαπάνες διοικητικές δαπάνες. Συχνά οι δαπάνες τους δεν είναι τέτοιου είδους. Αν, πάμε την, αν πάρουμε τον οργανισμό για τις χημικές ουσίες, δεν κάνουν διοικητική δουλειά. εφαρμόζουν ευρωπαϊκές πολιτικές και είμαστε πιο φθηνά από ότι αν κάνανε αυτή τη δουλειά τα κράτη-μέλη μόνο τους, το καθένα χωριστά. Ούτως ή άλλως, χάρη στην πρωτοβουλία του Κοινοβουλίου γίνεται αυτή η γενική εξέταση των οργανισμών. Γιατί θεωρήσαμε κάποια χρονική στιγμή ότι πολλαπλασιάζονται σαν μανιτάρια αυτοί οι οργανισμοί και ότι χρειαζόμαστε να έχουμε καλύτερο έλεγχο του κόστους που προκύπτει από αυτόν τον πολλαπλασιασμό. Η Γιούτα θα σας εξηγήσει ότι έχουμε φτάσει σε μια συνεννόηση με το Συμβούλιο για τους οργανισμούς. Δεν έχουμε νέα διαθεσμική συμφωνία, αλλά τέλος πάντων υπάρχουν κάποιες, κάποιες συμφωνίες σημαντική ίσως για το μέλλον των οργανισμών. Ειδικά αν εμεί στο Κοινοβούλιο χρησιμοποιήσουμε όπω πρέπει αυτή τη συμφωνία, αυτά τα λόγια, εν τα οποία, αυτέ τι διατυπώσει οποίε έχουμε συμφωνήσει, ούτω ώστε να αποφύγουμε τις πιο ανεπιθύμητες αποφάσεις που πήρε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, πούμε. Γιατί πολλές φορές χρειάστηκε η οργανισμοί αυτοί να αντιμετωπίσουν υψηλότερο κόστος ή διάφορες δυσκολίες που θα μπορούσαν να είχαν αποφευθεί. Η ερώτησή μου αφορά την προτάση της Κομισιόν. Η Κομισιόν μας εξήγησε ότι δεν σας αντιμετωπίζουν πιο σκληρά από ότι την Κομισιόν. Ότι μπορεί να υπάρχουν θέσεις που χειρεύουν σε κάποιους οργανισμούς, ότι μπορεί να υπάρχουν κάποια πλεονάσματα Δεν είναι δεδομένο ότι χρειάζεται και αυτές τις αυξήσεις κατά ανάγκη που αρχικά είχαν προβλεφθεί. Είπατε σύντομα ότι ήδη η πρόταση της Κομισιόν ήταν προβληματική. Μπορείτε να μας εξηγήσετε πιο συγκεκριμένα σε ποιο σημείο είναι προβληματική η πρόταση της Κομισιόν. Και γενικά πώς την ε, θεωρείτε. Είναι αποδεκτή. Καταλαβαίνω ότι έχετε πρόβλημα με τις περαιτέρω περικοπές προτείνει το Συμβούλιο. Δεύτερον, χάρη στην πρωτοβουλία της ειδική Επιτροπής, πάτε σε κάθε κοινοβουλευτική επιτροπή, συζητάτε στα πλαίσια ενός τακτικού διαλόγου, γνωρίζουν τη ε, δουλειά σας, ε, μαθαίνουν τα νέα καθήκοντα και τις αρμοδιότητες που σας φορτώνουν και οι δικευμένε επιτροπές είναι πολύ προσεκτικές. Ε, ξέρουν πολύ καλά ότι δεν μπορούν να αυξάνουν συνέχεια τον προπολογισμό, δεν μπορούν αιωνίως να προβλέπουν αυξήσεις. Από εκεί πρέπει να ξεκινήσετε ίσως. Θα ήθελα μια πιο λεπτομερή αξιολόγηση παρακαλώ της πρότασης της Κομισιόν πάντως. Ευχαριστώ, Άννα. Η Γιούτα. Ευχαριστώ. Ξέρουμε όλοι και το λέμε και ο ένας τον άλλον σε τέτοιες συνεδριάσεις πως οι υπηρεσίες αυτές κάνουν τη δουλειά αυτή, την εφαρμογή δηλαδή της ευρωπαϊκής πολιτικής και διοικητικά. Δηλαδή είναι, αν θέλετε, μια υπηρεσία η οποία ξελασπώνει, αν θέλετε, την Κομισιόν η οποία δεν θέλει να κάνει, ήδη θεωρεί ότι δεν μπορεί να κάνει κάποιες δουλειές. Αλλά βλέπουμε πως και στον προϋπολογισμό δεν γίνεται ποτέ λόγος για το ότι οι αποκεντρωμένες αυτές οι υπηρεσίες ανεξαρτήτως του είδους και της εργασίας τους ε, πάνε στην κατηγορία 5, δηλαδή στις διοικητικές δαπάνες. Όχι. Η Κομισιόν πάντα ήταν υπερήφανη να τηρεί το δικό της το κομμάτι μικρό, των διοικητικών δαπανών δηλαδή, και μετά έδωσε τη δουλειά της σε άλλες υπηρεσίες, αλλά δεν φαίνεται αυτό, γιατί φαίνεται κάπου στις λειτουργικές δαπάνες του προϋπολογισμού. Οπότε, εάν δεν ε, χρηματοδοτούνταν τουλάχιστον εν μέρη από τέλη, θα πήγαιναν από τα δικά μας εντός εισαγωγικών λειτουργικά έξοδα. Το ένα αυτό είναι το ένα. Αλλά και πάλι, να πω κάτι άλλο. Τελευταία φορά, στο πολιετέ δημοσιονομικό πλαίσιο του... Όταν παλέψαμε για το 2007-2013, κάποιοι βουλευτές είχαν την ιδέα όλες οι αποκεντρωμένες υπηρεσίε, να πάνε σε μία κατηγορία για να έχουμε μία καλύτερη ε, επίβλεψη των εξελίξεων κτλ. Η Κομισιόν αντιστάθηκε με νύχια και με δόντια. Όχι, αποκλείεται, δεν είναι δυνατόν, δεν πρέπει να υπάρχει πλαφόν κτλ. Καμία κατηγορία ποτέ. Εντάξει, οκ. Okay. Κάποιες από αυτές τις υπηρεσίες μετά βέβαια ήταν εναντίον, αλλά τώρα το κάνει απλά εντό της ε, διαδικασία του υπερπολογισμού και λέει θα πάνε όλα αυτά μαζί, παριστάνουμε σαν να ήταν μία κατηγορία και διοικητική μάλιστα και πρέπει να εξοικονομήσει 1% του προϋπολογισμού όπως κάνει και η Κομισιόν και όλοι οι υπόλοιποι, το κοινοβούλιο, δικαστήριο κτλ. κτλ. Όλοι πρέπει να εξοικονομήσουν 1%. Δεν είναι συνεπές αυτό, δεν είναι λογικό. Όταν το έμαθα και είδα πώς ήταν τα πράγματα, έγραψα μια επιστολή στον Επίτροπο τον κύριο Λεβαντόφσκι, δεν με ικανοποίησε η απάντηση, δεν ήταν σωστή η εξήγηση και δεν υπάρχει εξήγηση. Τι έχουμε εδώ πέρα. Αλλαγή της προηγούμενης πολιτικής δεν είναι ούτε λογικό ούτε συνεπές. Δεύτερον, πρέπει να γίνει συνολικά 1% εξοικονόμηση. Μα τι γίνεται με την αρχή που έχουμε πως νέα καθήκοντα σημαίνει νέα κονδύλια. Αυτό το λέμε ξανά και ξανά. Και πρέπει αυτό να ισχύσει κυρίως για τις αποκεντρωμένες αυτές τις που δεν έχουν και περιθώριο να κινηθούν εκτός του προπλογισμού τους. Και βεβαίω, εντάξει υπάρχει εν μέρη χρηματοδότηση από τέλη για κάποιους, αλλά ξέρω πως εδώ πέρα είναι οι λάθος άνθρωποι από την Κομισιόν, αλλά πρέπει να πει η Γενική ε, Διεύθυνση, να πει, ακούστε κύριοι, τα τέλη που εισπράττουμε τα θέμε για αυτή την πολιτική. Αλλά δεν μπορούν να το κάνουν. Γιατί Μα κάποτε πρέπει και οι υπηρεσίε αυτές με τα τέλη που εισπράττουν να πληρώσουν του ανθρώπου που κάνουν αυτή τη δουλειά. Το λέει και η Κομισιόν. Δεν μπορεί να δράσει σε ένα κενό. Εδώ πέρα πρέπει κάποτε και η Κομισιόν να παραδεχτεί πως δεν είναι δυνατόν κάποια πράγματα να γίνονται την τελευταία στιγμή. Και εμείς ε, πρέπει να δρούμε με αποθέματα, με μπλοκαρίσματα στη διαδικασία του προπολογισμού. Δεν είναι δυνατόν, είναι κουραστικό, είναι βαρετό. Ε, κάθε χρόνο στη διαδικασία του υπολογισμού έχουμε την ίδια δήλωση πως θέλουμε οι υπηρεσίες εκείνες οι οποίες χρηματοδοτούνται εν μέρη από τέλη να έχουν την δυνατότητα με τα έσοδα αυτά να κάνουν κάτι ε, σε αντίθεση με τις άλλες οι οποίες εξαρτώνται 100% από τον κοινοτικό προβληματισμό γιατί αυτή είναι η διαφορά. Δεν μπορούν να εξυπηρετήσουν την ε, βιομηχανία και όποιον άλλον πληρώνει τέλη και να ξεκινάνε κάθε χρόνο από το μηδέν και να μην υπάρχει κανένα πλεόνασμα, να μην μεταφέρεται τίποτα κτλ. Υπάρχουν ε, πολλές από αυτέ τι υπηρεσίε οι οποίες θα είχαν κάποια μεγαλύτερη ευελιξία για την διοίκηση του προπολογισμού τους με αυτά τα τέλη. Και τώρα προστίθεται σε όλα αυτά. Και δεν μου δώσατε απάντηση εδώ. Θέλω να μάθω τι κάνετε μαζί μας για να πούμε στο Συμβούλιο δεν πάει άλλο αυτή η κατάσταση. Πήρατε το 1% και ξανά Στι υπηρεσίες την πέφτατε. Τι κάνετε εκεί πέρα δηλαδή. Το Συμβούλιο εννοώ τι κάνει. Bien. Madame la vice-présidente. Η αντιπρόεδρος, η, εισηγήτρια ειδικευμένη, εξειδικευμένη στους οργανισμούς έθεσε ορισμένα μεγάλα ερωτήματα. Μερικές παρατηρήσεις. Συγγνώμη, συγγνώμη. Ντομινίκ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. ο οποίος έχει δεσμούς με την Βαλανσιά, την πόλη Βαλανσιά, κατά συνέπεια και με έναν οργανισμό. Εντάξει, με ξεσκέπασες. Λοιπόν, ε, δεν θα συνηγορήσω μου, αλλά θα κάνω μερικές ε, παρατηρήσεις. Εδώ έχουμε το 35% του προσωπικού της πόλης της Μασαλίας. Δεν νομίζω ότι η συζήτηση είναι δημοσιονομική συζήτηση. Γι' αυτό λοιπόν ε, χανόμαστε κιόλας όταν συζητάμε με το Συμβούλιο. Οι οργανισμοί τι είναι. Είναι ένα μέσο που μας επιτρέπουν να εξομαλύνουμε και να εφαρμόσουμε τις κοινωνικές διατάξεις. Εργάζονται για τη λειτουργία και την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση. Όποιος και να είναι ο τομέας τους. Και ποιος προτείνει στο Συμβούλιο τον προϋπολογισμό για τους οργανισμούς, μα υπάλληλοι εθνικών υπουργείων Άτομα δηλαδή τα οποία μπορούν να αισθάνονται ε, ότι απειλούνται ε, μέσω των οργανισμών ε, ή αισθάνονται να απειλούνται γενικά. Είναι ανταγωνιστές λοιπόν. Αυτοί οι ανταγωνιστές ορίζουν τον προϋπολογισμό. Οι οργανισμοί είναι το σύμβολο του, Ευρωπα... του του ευρωπαϊκού όπλου είναι το λειτουργικό πεδίο της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης. Και σίγουρα τα προσχήματα είναι δημοσιονομικά. Για... Και καταλαβαίνουμε γιατί είναι ηλίθια αυτά τα μέτρα, λέει ο μιλητής, άμα λάβουμε υπόψη όσα μας είπε και η αντιπρόεδρος. Λοιπόν, η μέθοδος είναι ηλίθια το να παίρνει κανείς ένα τσουβάλι όλους τους οργανισμούς χωρίς να βλέπει αρμοδιότητες κτλ. Απλά και μόνο εδώ έχουμε ένα σαφές πεδίο, την, την εικόνα ενός σαφούς πεδίου μεταξύ διακυβερνητικής και κοινοτικής μεθόδου. Υπάρχει το κοινοβούλιο και οι Κομισιόν που, θέλ, που παίζουν το ρόλο της, της ευρωπαϊκής πολιτικής. Λοιπόν, θα ήταν ε, το μυστήριο της Πουλτσινέλα να μην δούμε ότι το Συμβούλιο είναι αυτό διακυβερνητική. Λοιπόν, στα γαλλικά θα λέγαμε Λάγκ de σίκα σίκα σκάφη σκάφη». Δεν, είναι Λάγκ de Σύμφωνο. Η Κομισιόν υπέβαλε προτάσεις που μπορεί να φαίνονται σκληρές στους οργανισμούς αλλά μπορούν να εξηγούνται και από το λόγο ότι και η ίδια η Κομισιόν επέβαλε στον εαυτό της ε, λιτότητα ως προς τις δαπάνες λειτουργίας στον προπολογισμό 2013. Και αυτό πρέπει να το έχουμε στο νου μας. Στις ε, θέσεις που έχει λάβει το Συμβούλιο σε επίπεδο Κορεπέρ, έτσι όπως υπόθηκε. Διότι πρόκειται για λερναία ύδρα το Συμβούλιο, με, με πάρα πολλά πλοκάμια, χιλιάδες πλοκάμια. που λαμβάνει αποφάσεις αντιφατικές μεταξύ τους, ανάλογα με τη στιγμή, με τη φύση των συμβουλίων, με το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Μα είναι απίθανο, αδιανόητο. Μετά από το τελευταίο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, γιατί μίλησαμε πολύ για τον προπολογισμό και σήμερα το πρωί. Μετά το τελευταίο Συμβούλιο της 28ης-29ης Ιουνίου, όπου το Συμβούλιο επίσημα αποφασίζει να ενισχύσει την δημοσιονομική εποπτεία για να καταλήξουμε στην τραπεζική ενότητα. Πέντε μέρες μετά η Κορεπέρ μειώνει τις πιστώσεις των τριών οργανισμών εποπτείας που συστάθηκαν πέρσι και που δεν είχαν δηλαδή και τους ε, κατάλληλους πόρους, δεν πέτυχαν να τους έχουν, παρά μόνο χάρη του, χάρη του Κοινοβουλίου και της Επιτροπής Προϋπολογισμών. Το 2012 εμείς επιμείναμε να αποκαταστήσουμε τα κονδύλια τα οποία είχε ζητήσει η Κομισιόν για αυτούς τους οργανισμούς και το Συμβούλιο είχε μειώσει. Είναι παράλογο, είναι απίθανο. Επίσης, στη διάρκεια της χρονιάς διαπιστώσαμε και άλλες αντιφάσεις. Ένα άλλο συμβούλιο, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, είχε ζητήσει να ενισχύσουμε τον έλεγχο στα εξωτερικά σύνορα και αναθεώρηση του, του Σέγγεν. Και την άλλη, την επόμενη εβδομάδα η Κορεπέρ μείωνε τα κονδύλια της Frontex. Ε, όλα αυτά είναι ε, ασυναφή. Και όπως το position paper το οποίο μας εστάλει λέγεται λαμπρά, μας το είπε ο Διευθυντής Πρόεδρος της Τρόικα, βλέπουμε ότι αυτοί οι οργανισμοί είναι μικροί οργανισμοί και χρειάζονται κριτική μάζα διότι κάτω από ένα επίπεδο δεν έχουν καμία ευκαιρία επιτυχίας όταν πρόκειται δηλαδή για επιβολή κανόνων σε ένα χώρο με 500 εκατομμύρια κατοίκους. Διατρέχουμε τον κίνδυνο η δουλειά να είναι κακοφτιαγμένη, όπως επίσης και επανέρχομαι διότι ο Ντομινίκ ε, ε, Ρίκε μπήκε στο ψαχνό της υπόθεσης όλα αυτά να στοιχήσουν πολύ πιο ακριβά. Διότι οι ευρωπαϊκοί οργανισμοί μη έχοντας τα απαραίτητα κονδύλια δεν κάνουν σωστή δουλειά, οπότε μία, ένας ήδη υπάρχον εθνικός οργανισμός κάνει τη δουλειά στη θέση του ευρωπαϊκού οργανισμού με αυξημένα κονδύλια ή αν δεν υπάρχει αυτός ο οργανισμός σε εθνικό επίπεδο δημιουργείται διότι οι Βρυξέλλες θεωρούνται ανίκανες. Επιμένω λοιπόν εγώ σε ένα θέμα το οποίο δεν ενδιαφέρει καμία κυβέρνηση πουθενά και κανέναν υπουργό οικονομικών και δεν ενδιαφέρει ούτε το Ευρωπαϊκό Ελεγκτικό Συνέδριο, δυστυχώς ελπίζω κάποιος να είναι εδώ, να τα ακούσει, ούτε τους, τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια. Υπάρχει λοιπόν ένα θέμα επικάλυψης μεταξύ εθνικών και ευρωπαϊκών διοικήσεων και Και όταν μεταφέρουμε αρμοδιότητες από εθνικό επίπεδο σε ευρωπαϊκό επίπεδο, θα πρέπει να θέτουμε την απέτηση της αντίστοιχης μείωσης των κονδυλίων, των διοικητικών κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο, ούτως ώστε η ευρωπαϊκή οικοδόμηση και η κατανομή αρμοδιοτήτων μεταξύ εθνικού και ευρωπαϊκού επίπεδου να γίνεται με σταθερές δαπάνες και όχι αυξάνοντας συνολικά την γραφειοκρατία. Και οι υπουργοί αντί να λένε θαύμα, τι ωραία, η Ευρώπη θα είναι τώρα αρμόδια για την ασφάλεια στα τροφίμων ή για την αεροπορική ασφάλεια κλπ. κλπ. Αντί να λένε αυτό και, και μειώνω τους εθνικούς μου υπαλλήλους, τι δεν λένε τίποτα. Τώρα δημόσια είμαστε εδώ και το λέω και δημόσια δηλαδή. Η χώρα μου η Γαλλία εφάρμοσε το Σέγγεν το 1993, δηλαδή τέρμα η τελωνιακή έλεγχη μέσα στην Ένωση, κατάργηση των αστυνομικών ελέγχων μέσα στο, για, για τα φυσικά πρόσωπα μέσα στον ευρωπαϊκό χώρο. Όταν, όταν έγινε υπουργό ε, Δήμου Οικονομικών μετά από δύο χρόνια, τι διαπίστωσα ότι είχαν αυξήσει τον αριθμό των τελωνιακών, των Γάλλων τελωνιακών, δύο, στα δύο χρόνια τις ε, διακοπ... της ε, σε ισχύ στο Σέγγεν. Γιατί, για να παρηγορήσουν τους τελωνιακούς ότι δεν είχαν πια δουλειά. Λοιπόν, βέβαια ξέρετε υπάρχουν χώρες οι οποίες τις οποίες τις διαχειρίζονται καλύτερα από τη δικιά μου. Αλλά αν ήμασταν σοβαροί και οι ηγέτες μας είναι σοβαροί και πραγματικά θέλουν το value for money, θα έπρεπε να αντικαταστήσουν όλη την αστυνομία που ασχολείται με τον έλεγχο στα σύνορα, χερσαία ή ε, διαέρος με το Frontex. Αλλά δεν γίνεται τέτοιο πράγμα. Αυτό το οποίο κάνει το Συμβούλιο υπό το πνεύμα που μας ανέφερε ο κύριος ε, Ρικέ είναι να μειώνουν την Ευρώπη θεωρώντας ότι η ευρωπαϊκή διοίκηση είναι ένας επικίνδυνος ανταγωνιστής. Τώρα, αυτό το οποίο συνειδητοποιούμε είναι ότι οι οργανισμοί μέτρησα εγώ 33 συν 4 ακαθορίστου φύλου. Δηλαδή έχουμε 4 τρανσεξουέλ, λέει ο πρόεδρος. Πώς... Τέσσερις φιλομεταβατικοί λοιπόν, ή ορφανοί όπως θέλετε, Αλλά και η Κομισιόν έναντι αυτών των 33 και 4 έχει την ίδια στάση πολλές φορές με τα κράτη-μέλη. Αγαπάει με τους οργανισμούς της, αλλά υπάρχουν γενικές διευθύνσεις οι οποίες ε, εμπίπτουν στον πειρασμό να κρατήσουν το μάξιμουμ των εξουσιών στο Μπέρλεμον και να μην πρικοδοτούν έπαρκος τους εξωτερικούς οργανισμούς ανά την Ευρώπη. Είναι, ορφανές είναι ορφανή πολιτικά οι οργανισμοί. Και αυτό που θέλω να πω στους τρεις διευθυντές της Τρόικα Λοιπόν, τα μέσα δεν είναι ατελείωτα. Να ξέρετε, εδώ έχετε έναν πατέρα και μία μητέρα, ορίστε, τη Γιούτα. Τα μέσα δεν έχουν εξαντληθεί. Αλλά εμείς δεν θέσουμε το πρόβλημα, όπως το έκανε και η Γιούτα, όπως το είπε και ο Ντομινίκ Η δημοσιονομική πρόκληση δεν είναι τόσο σοβαρή. Πολιτική είναι η πρόκληση. Ο Σαλβαδόρ. Για τους τρεις οργανισμούς εποπτείας, τον έναν εποπτεία, τραπεζικής εποπτείας και τους άλλους δύο, διαπίστωσα ότι έχουμε την ίδια ανησυχία από το 2012 και κάτι πολύ συγκεκριμένο που αφορά στην αξιολόγηση των πόρων αυτών των οργανισμών. Η Κομισιόν τους αξιολογεί διαφορετικά από τους άλλους οργανισμούς και, η εκτίμηση των, και έχουμε μία εκτίμηση των απαραίτητων θέσεων που δεν ανταποκρίνεται με το establishment plan που έχουν ορίσει οι οργανισμοί και υπάρχει λοιπόν μία ασυμβατότητα μεταξύ αυτών, αυτής της καταγραφής των θέσεων. Θα έπρεπε να υπάρχει μια μεγαλύτερη συμφωνία μεταξύ μεγαλυτερη συμφωνια μεταξυ κομισιών και των οργανισμών όταν θεσπίζουν το οργανόγραμμά τους και για την εποπτεία ε, για τον οργανισμό για την εποπτεία ξέρετε το κοινοβούλιο έπαιξε σημαντικό ρόλο διότι ε, για μας είναι σημαντικότατο πολιτικά και θα έχει τον ίδιο προπολογισμό με πέρσι αλλά εμένα μου φαίνεται παράλογο το επαναλαμβάνω να υπάρχουν αυτές οι ανισότητες μεταξύ της εκτίμησης των απαραίτητων πόρων που προβλέπει η Κομισιόν και των προβλέψεων των οργανισμών. Θα χρειαζόταν ένας διάλογος μεταξύ όλων αυτών. Ευχαριστώ. Κύριε Διευθυντά, θέλετε να ξαναπάρει το λόγο για να απαντήσετε σε κάποιες παρατηρήσεις των συναδέλφων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Νομίζω πως παρατηρήσεις των βουλευτών είναι θετικές. Γιατί γεγονός είναι πως σε τελική ανάλυση δεν έχουν φωνή οι αποκεντρωμένες υπηρεσίε ε, για ζητήματα για να εκθέσουν ε, τα επιχειρηματά τους γιατί ακόμα πράγματα τα οποία στο χαρτί φαίνονται λογικά αλλά αν δει κανεί την πραγματικότητα υπάρχουν ε, πράγματα που δεν στέκουν. Να φέρω ένα παράδειγμα από τη δική μου υπηρεσία. Για τα βιοκτώνα. Είναι μια δουλειά την οποία πριν έκανε η Κομισιόν. Μας μεταφέρει λοιπόν η Κομισιόν τη δουλειά τη, χωρίς να μα ρωτήσει κιόλα. και λέει μετά, α, δεν θα λάβετε όμω και τι θέσει που σας υποσχεθήκαμε, Έχουμε μια ανομαλία εδώ πέρα λοιπόν. Δηλαδή εφενός έπρεπε να περικόψουν τις δικές τους θέσεις εφόσον ε, δίνουν τις αρμοδιότητες και δεύτερον εάν ζητάνε από μια υπηρεσία να κάνει αυτό το οποίο έκαναν οι ίδιοι πριν να έχει τους απαραίτητους σπόρους. Ένα παράδειγμα σας δίνω. Και είμαι σίγουρος πως το ίδιο συμβαίνει και αλλού. Έχουν νέα καθήκοντα τα οποία δεν είναι υποχρεωτικό ότι ζήτησαν και απογοητεύονται γιατί ε, δεν θα είναι σε θέση να τα επιτελέσουν σωστά ενώ ο πολίτης αναμένει βεβαίως αποτελεσματική λειτουργία. Αυτό ήθελα να σας πω ως παράδειγμα και είμαι σίγουρος πως ε, και οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες που μόλις αναφέρθηκαν, οι τρεις αυτές, ε, δυσκολεύονται και έχουν οπωσδήποτε πολύ δύσκολα καθήκοντα στην οικονομική κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε και χωρίς τους κατάλληλους πόρους είναι αδύνατον να συνεισφέρουν αυτό το οποίο πρέπει για να βοηθήσουν ε, την Ευρωπαϊκή Ένωση να βγει από το χάλι στο οποίο βρίσκεται αυτή τη στιγμή. Από οικονομική σκοπιάς. Οπότε ζητάμε από την Κομισιόν να βοηθήσει τι αποκεντρωμένες αυτέ τι υπηρεσίε μαζί με το Κοινοβούλιο να αποκαταστήσει αυτά τα λάθη και όπου είναι αυτό δυνατόν να διορθώσει την κατάσταση, να διορθώσει τα λάθη του Συμβουλίου δηλαδή. Σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Διευθυντά. Να υπενθυμίσω ότι έχουμε και μια ομάδα εργασίας εδώ και λίγο καιρό, διαθεσμικού χαρακτήρα, που παρακολουθεί το έργο των οργανισμών. Θέλω να τιμήσω εδώ την Γιούτα και τον Γιάνσεν, την κυρία Γκρέσλε επίσης που μας εκπροσωπούν και παίζουν ενεργό ρόλο και να υπενθυμίσω ότι αυτή η ομάδα στις 5 Ιουλίου έστειλε στη διάσκεψη των Προέδρων την κοινή δήλωση για τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και οργανισμούς που εγκρίθηκε από τη διάσκεψη. Πού είναι ο μπούσουλάς μας στις σχέσεις με τους οργανισμούς και ο μπούσουλάς μας για την προετοιμασία των αποφάσεων που λαμβάνονται για τις υπηρεσίες, ιδίως για τα δημοσιονομικά θέματα. Ε, είναι ο καρπός τριών χρόνων εργασίας. Η Ευρώπη χτίζεται με πολύ υπομονή. Ευχαριστώ. Κλείνω αυτή τη συζήτηση. Ευχαριστώ ακόμα τους τρεις διευθυντές της Τρόικα και τους άλλους διευθυντές που είναι μέλη εκπρόσωποι των οργανισμών που είναι παρόντες εδώ στη συζήτηση. Τους διαβεβαιώνω ότι θα έχουν την υποστήριξή μας. Συνάδελφοι, τώρα συνεχίζουμε τις εργασίες μας για τις εκθέσεις. Ο Ντομινίκ Ρικέ είναι σε φόρμα. Του προτείνω να μας παρουσιάσει την έκθεσή του για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, το σημείο 17 της Μέσης Διάδαξης. Ντομινίκ, στο λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω ότι στο νέο πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο η Κομισιόν παρουσίασε ένα σύνολο προτάσεων πρωτοβουλία με σκοπό να πλουστεύσουμε τον τρόπο χρηματοδότηση των εσωτερικών του κλάδου των εσωτερικών υποθέσεων. Η χρηματοδότηση αυτή θα κατανεμηθεί σε δύο ταμεία, ένα για το άσυλο και τη μετανάστευση, δεν είναι αυτό που θα μας απασχολεί σήμερα, και ένα ταμείο για την εσωτερική ασφάλεια που διαιρείται σε δύο μέσα αυτό. Το πρώτο αφορά την ε, ασφάλεια των εξωτερικών συνόρων και το δεύτερο που είναι και το αντικείμενο της σημερινής έκθεσης αφορά την αστυνομική συνεργασία, την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος καθώς και τη διαχείριση των κρίσεων. Το να πούμε ότι μια και οι διαπραγματεύσεις για το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο 2014-2020 είναι αυτές που είναι, δεν θέλω να το σχολιάσω αυτό, γιατί εντάξει, αν είναι μια επιτροπή που τα ξέρει αυτά τα θέματα, είναι αυτή εδώ η επιτροπή. Ε, έχουμε λοιπόν το πλαίσιο αυτό ε, στον κανονισμό, αλλά δεν πρόκειται να καθοριστεί αυτό οριστικά πριν από μια συνολική συμφωνία. Και τα νούμερα όλα αυτά να τα δείτε εντό αγγυλών. Θα δούμε τι θα απογίνουν τελικά. Ούτω ή άλλω αυτό συνδέεται και με το θέμα των οργανισμών για το οποίο μόλι συζητήσαμε. Το πεδίο εφαρμογή λοιπόν αυτού του μέσου είναι αρκετά ευρύ γιατί ε, περιλαμβάνει την, το συντονισμό και την ανταλλαγή καλών πρακτικών μεταξύ των αστυνομικών αρχών των κρατών μελών τις δραστηριότητες αξιολόγησης, ανάλυσης και εποπτείας, τις δράσεις ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης, την κατάρτιση του προσωπικού, την αγορά και τη δοκιμή νέου εξοπλισμού και υλικού. Προβλέπει επίσης ενδεχομένως τη συμμετοχή των τρίτων χωρών ή κάποιων τρίτων χωρών σε υπό κάποιους όρους. Το δυνητικό ποσό ε, στα πλαίσια του πολιτού πλαισίου αν θυμάμαι καλά, και το βάζοντα αγγελών, είναι 1,128 δις ευρώ. Τα μισά ε, τη χάνουν κεντρική διαχείριση και αυτό είναι καινοφανέ στοιχείο σε σχέση με το προηγούμενο ταμείο ε, και το μισό θα πάει στη διαχείριση των κρατών μελών υπό την αιγίδα και τον έλεγχο της Επιτροπής. Δηλαδή, επιμερισμένη διαχείριση και έλεγχος. Ο εισηγητής σας υποστηρίζει αυτή την πρόταση που είναι μια πρόταση και απλούστευσης αλλά και εξορθολογισμού ταυτόχρονα. Δεν θα κάνω σχόλια στο δημοσιονομικό κονδύλι, λαμβάνοντα υπόψη όλα όσα ακούσαμε μέχρι στιγμή. Από ό,τι φαίνεται είναι αρκετά προσαρμοσμένο. Δεν φαίνεται να τα έχουν χάσει εδώ οι θύνοντε. Κάποιε τροπολογίε θα πρέπει να γίνουν παρόλα αυτά και θα αφορούν ουσιαστικά τον έλεγχο, το δημοκρατικό έλεγχο των δαπανών είναι ένα θέμα που η δική μας Κοινοβουλευτική Επιτροπή είναι πολύ ευαισθητοποιημένη. Η προσπελασιμότητα των προγραμμάτων για όλους τους συμμετέχοντες, η διαφάνεια των δημοσιονομικών πόρων και μια επαρκής παρακολούθηση είναι πάντα θέμα με τα χρηματοδοτικά μέσα αυτό. τα αποτελέσματα και η ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία επίσης είναι ένα θέμα που μας απασχολεί πολύ εμάς και συχνά είναι απόν στα θέματα ασφάλειας και η ορατότητα των δράσεων της Ένωσης. Μετά από την επιμερισμένη διαχείριση που αποφασίστηκε, θα πρέπει να υπάρχει αποτελεσματικό συντονισμό ε, μεταξύ τη Ένωση και των κρατών μελών. Γιατί τα μισά πηγαίνουν σε κεντρική διαχείριση και τα μισά σε επιμερισμένη διαχείριση. Άρα θα πρέπει να είναι συντονισμό για τα ίδια θέματα αυτών των δύο ειδών διαχείριση. Έχω υπόψη μου δηλαδή να είμαστε σίγουροι τόσο ώστε η ευθυγράμμιση των εθνικών προγραμμάτων να γίνεται ε, μέσα στα πλαίσια τη Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Εσωτερική Ασφάλεια τη Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα θέλαμε αυτό το μέσο να επανεθνικοποιηθεί δηλαδή, κάτι που θα ήταν καταστροφικό. Γι' αυτό λοιπόν θέλω να τονίσω ότι η κεντρική διαχείριση θα πρέπει να είναι ο κανόνας, έτσι. Θα ήταν πιο προσήκον. Γίνεται μια συζήτηση γύρω από αυτό. Η δράση των κρατών μελών θα πρέπει τουλάχιστον να θεωρείται συμπληρωματική. Για τα εθνικά ποσά τώρα, προτείνω να βάλουμε ένα κριτήριο που δεν υπάρχει. Υπάρχουν κάποια κριτήρια πληθυσμού, ε, επιφάνειας, ε, ακαθάριστου εθνικού προϊόντος, ε, στρατηγικών υποδομών, αλλά λείπει και το ποσοστό εγκληματικότητα, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Γιατί είναι ένα από τα στοιχεία που καθιστά απαραίτητη την χρήση του μέσου στην κάθε επικράτη του κράτους μέλους. Τώρα, Θέλω να τονίσω τη δυνατότητα συνεργασίας με τη Europol και να κάνουμε κάποιες τροπολογίες τον Αύγουστο. Ξεχάσαμε την, το λαθρεμπόριο προστατευόμενων ειδών στον κατάλογο αυτών των ε, υποαπειλή ειδών. Και τέλος, είμαι έτοιμος να απαντήσω σε όλες τις ερωτήσεις σας για αυτή την γνωμοδότηση και να συνεχίσω τη συνεργασία με τους συναδέλφους και τους εισηγητές, τους κοιόδης εννοείται. Αυτά, Πρόεδρε, σε ό,τι αυτή την έκθεση που θα καταθέσω. Ευχαριστώ, Ντομινίκ. Σχόλια παρατηρήσεις. Όχι. Αυτή η έκθεση, λοιπόν, είναι τμήμα μια ομάδα τεσσάρων εκθέσεων, όπως είπε και ο Ντομινίκ Ρικέ, για τη χρηματοδότηση της πολιτικής εσωτερικής ασφάλειας, ασύλου, προστασίας των συνόρων και το χρονοδιάγραμμα για αυτή την έκθεση είναι το ίδιο. Η καθήλυνα αρμόδια επιτροπή είναι η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ, εμείς νομοδοτούμε απλώς. Μετά την ανταλλαγή απόψεων σήμερα, η προθεσμία για τις τροπολογίες είναι η 19η Ιουλίου θα πρέπει να ψηφίσουμε την γνωμοδότησή μας στις 6 Σεπτεμβρίου στην επόμενη συνεδρίαση της Επιτροπής μας και η Λίμπε από πλευρά της θα υιοθετήσει το κείμενό της το Νοέμβριο. Όλα αυτά είναι σε ένα σωστό πλαίσιο με τη θέλησή μας να περάσει το κείμενο αυτό ε, στην Ολομέλεια μέχρι το τέλος του 12. Ευχαριστώ τον Ντομινίκ Χρικέ. Τώρα οι άλλες τρεις εκθέσεις για τα συναφή θέματα είναι θέματα της Μόνικα αλλά δεν είναι εδώ. Προτείνω λοιπόν να περάσουμε στο σημείο 7 της Helga Τριπέλ για ένα θέμα που μας είναι πολύτιμο, που είναι ε, η δράση για το πρόγραμμα LIFE. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, όπως και η συνάδελφός μου εδώ εξεβονίμων. Είμαι και εγώ κουρασμένη. Εγώ θα προσπαθήσω να είμαι σύντομη. από την υποβάθμιση του περιβάλλοντος και την κλιματική αλλαγή έχουμε κάποιες πολύ σοβαρές αλλαγές που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση όπως όλοι ξέρουμε και όπως συνεχώς επαναλαμβάνουμε με τα μεγάλα μας ψηφίσματα στην Ολομέλεια και στην Επιτροπή Καταπολέμησης Κλιματικής Αλλαγής και το να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση στον κίνδυνο που συνδέεται με αυτήν πρέπει να είναι μια προτεραιότητα των πολιτικών μας προσπαθειών. Όπως εκφράζεται η στρατηγική της Ευρώπης 2020 υπάρχει επίγουσα ανάγκη για πιο αποφασιστική πολιτική δράση. Και άρα θα ήθελα να σας υπενθυμίσω πως όταν θα ψηφίσουμε την έκθεση ΣΟΥΡ, όταν ψηφίσαμε την έκθεση ΣΟΥΡ, με συγχωρείτε, τον Ιούλιο του 2011, τονίσαμε την σημασία ενός ξεχωριστού χρηματοδοτικού μέσου για το περιβάλλον και το κλίμα. Έχουμε δηλαδή εδώ πέρα την ραχοκοκαλιά των προσπαθειών διαφύλαξη του περιβάλλοντος με πάρα πολύ μικρές επενδύσεις στα οικολογικά και κοινωνικά ωφέλη ανταποκρίνονται σε πολλούς στόχου τη Ευρωπαϊκής Ένωσης όμως το πρόγραμμα LIFE είναι 0,23% του ε, πουδοπού 2007-2013 πολύ περιορισμένο ποσό χρημάτων και άρα αυτό το οποίο προτείνω είναι να αυξήσουμε το ποσοστό στον προπολογισμό σε 0,5%. Ξέρω πως υπάρχουν ΜΚΟ που θέλουν να πάνε ακόμα και παραπέρα. Αλλά θεωρώ πως εάν έχουμε την πολιτική δέσμευση να διπλασιάσουμε το ποσοστό του προγράμματος Life με όλα τα προβλήματα που έχει ο προϋπολογισμός νομίζω πως είναι ήδη κάτι φιλόδοξο και γνωρίζουμε και νομίζω πως ε, και από πολιτική σκοπιά είναι πάρα πολύ σημαντικό τα έργα του LIFE ε, αποδίδουν οικονομικά, εξασφαλίζουν θέσεις εργασίας και αποδίδουν και καινοτόμα έργα σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα αναφέρω κάποια πράγματα για να σας υπενθυμίσω αφορώ την αποθήκευση του άνθρακα σε δίκτυα του Natura 2000. Μιλάμε για 9,6 δισεκατομμύρια τόνους άνθρακα την περίοδο που μας πέρασε. Παραδείγματο χάρη, οι επισκέπτες των ε, περιοχών Natura Μιλάμε για 1,2 έως 2,2 εκατομμύρια επισκεπτών την ημέρα, οι οποίοι επωφελήθηκαν ε, σε ένα ποσό το οποίο υπολογίζεται από 50 έως 85 δισεκατομμύρια ευρώ. Υπάρχουν λοιπόν περιβαλλοντικές πτυχές από την αναζωογόνηση της φύσης και είναι και μια επένδυση η οποία δημιουργεί βεβαίως ε, λεφτά. Είναι ένας πολύ καλός συνδυασμό. Και υπάρχουν και πολύ καλά παραδείγματα στα κράτη-μέλη για το ότι το οικοσύστημα υποφελείται από την αποκατάσταση της φύσης και μετά από τη σύνοδο του Ρίο συν 20 αυτό νομίζω είναι σημαντικό να το ξαναπούμε αλλά είχαμε και δημιουργία θέσεων εργασία μέσω της αποκατάστασης οικοσυστημάτων δουλειέ σε ανθρώπου οι οποίοι ήταν άνεργοι για πολύ καιρό οπότε έχουμε και κοινωνική πτυχή τόσο δεν θέλω να τα αναφέρω όλα αλλά έχουμε ένα καλό συνδυασμό οικολογικής, οικονομικής και κοινωνικής προσέγγισης και ωφέλους. Είπα ήδη πως πρέπει να αυξήσουμε το ποσοστό του προϋπολογισμού στο 0,5% και μετά νομίζω πως είναι σημαντικό μια τροπολογία μου να έχουμε ένα ποσό το οποίο δεν θα είναι χαμηλότερο από το 0,37% του συνολικού φακέλου που θα πρέπει να πάει στο υποπρόγραμμα περιβάλλον το άλλο υποπρόγραμμα είναι του κλίματος και αυτό πρέπει να είναι 0,125%. Αυξημένος αριθμός ειδών έργων, δηλαδή εισαγωγή ολοκληρωμένων έργων που έχουμε στη νέα πρόταση, δεν πρέπει να μας οδηγήσει σε αντικατάσταση υφισταμένων επιτυχών έργων. Γιατί αν θέλουμε να συνδυάσουμε παλαιά και νέα έργα, δεν είμαι κατά. Αλλά αυτό σημαίνει πως θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την παλαιά προσέγγιση και όπως είπα η συνέπεια είναι η αύξηση του προϋπολογισμού στο 0,5%. Για το ζήτημα της συγχρηματοδότησης, ε, το μέγιστο ποσοστό συγχρηματοδότησης δεν θα υπερβεί το 50% κατά κανόνα. Αλλά για μένα, για πολιτικούς λόγους δεδομένης της κρίσης, είναι σημαντικό να υπάρχει η πιθανότητα για κάποιες χώρες και λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες και κράτη-μέλη με προσωρινές δυσκολίες να είναι επιλέξιμα για μια συγχρηματοδότηση μέχρι και 75% γιατί αυτό σχετίζεται με την όλη πολιτική επικοινωνία. Τι μπορούμε να κάνουμε γρήγορα για να βοηθήσουμε περιφέρειες και κράτη-μέλη με δυσκολίες και άρα χρειάζεται μια κάποια ευελιξία. Έχουμε σα, σαφείς αρχές όσον αφορά το ποστό χρηματοδότησης. Αλλά σε κάποιες περιπτώσεις ε, πρέπει να πάμε ακόμα παραπέρα. Μετά πρέπει να δούμε το τι θα κάνουμε με τον ΦΠΑ. Και εδώ πέρα πρέπει να έχουμε ένα ευέλικτο σύστημα. Κανονικά ο ΦΠΑ δεν είναι επιλέξιμη δαπάνη αλλά αν υπάρχουν ειδικέ ανάγκες πρέπει να υπάρχει δυνατότητα να τις αντιμετωπίσουμε. Θα μείνω σε αυτό, λοιπόν. Ελπίζω να δείτε τις προτάσεις μου και ελπίζω να επιτύχουμε περισσότερα με το πρόγραμμα αυτό και νομίζω πως έχει αποδειχθεί πως είναι ένα καλό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με πολλές επιτυχίες και πρέπει άρα να το συνεχίσουμε. Ευχαριστώ. Γιούτα. Ε, ευχαριστώ. Θέλω σύντομα να αναφερθώ στην έκθεση της Χέλγας. Πράγματι το πρόγραμμα LIFE είναι από τα πιο επιτυχή, εάν όχι το επιτυχέστερο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εντάξει και το Εράσμους καλό είναι εντάξει. Αλλά το LIFE ε, για μένα έχει πιο γρήγορα και μετρήσιμα αποτελέσματα. Όλα αυτά τα οποία είπε η Χέλγα τα υποστηρίζω και πρέπει να πω, να προσθέσω, το είπα και χθες, στη δική μου ομάδα εργασίας του προπολογισμού και τώρα το λέω σε όλους τους συναδέλφους. Εγώ είμαι η σκιώδη συγγήτρια εδώ για το Σοσιαλδημοκράτη. Είμαι η συγγήτρια στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και στηρίζω κάθε μία τροπολογία της Χέλγκας Δηλαδή, αν μπορούσα εγώ να κάνω τον κατάλογο των ψηφοφοριών χωρίς κανέναν από τους συναδέλφους από την ομάδα μου, θα έβαζα παντού ένα συν. Και για το 0,5%. Οπωσδήποτε μας κάνουν λόμπι οι περιβαλλοντικές οργανώσεις που λένε ούτε το 0,5 δεν φτάνει. 1% τουλάχιστον. Και ε, δεν είναι μυστικό, το ξέρετε. Και η Γερμανική Βουλή ακόμα αποφάσισε με, πως 0,7% του προπολογισμού θα πρέπει να πάει για το ΛΑΙΦ. Αλλά ξέρουμε πως ε, τα πράγματα είναι όπως και στο Συμβούλιο. Δεν ξέρει η αριστερά τους τι πει η δεξιά τους εκεί μέσα. Ε, οπότε αυτό δεν είναι το μέτρο της καλής βούλης των Εθνικών Κοινοβουλίων, αν θέλετε. Το 0,5 είναι ρεαλιστικό. Δεν είναι στο, στην, δεν έχει φτάσει στο ταβάνι. Πατάμε γεραστική και θέλουμε να προχωρήσουμε προς τα μπρος. Ε, είπα και σε άλλο πλαίσιο πως πρέπει να ακολουθήσουμε την αρχή νέες αρμοδιότητες, νέα κονδύλια. Γι' αυτό χρειάζεται η αύξηση. Στο παρελθόν είχαμε πολύ επιτυχή προγράμματα βιοπικιλότητας με το Natura 2000, με το Life κτλ. Τώρα προστίθεται, κάτι το οποίο είναι σωστό, η προστασία του κλίματος. Και χρειάζεται περισσότερα λεφτά. Και επιπλέον υπάρχει υπάρχουν αυτά τα ολοκληρωμένα έργα, τα νέου τύπου, όπου μετά ε, το live ε, από εκεί πέρα θα χρηματοδοτεί ένα μικρό κομμάτι και το υπόλοιπο κομμάτι θα πάει από τα μεγάλα ας πούμε ταμεία. Λογικό αυτό, σωστή προσέγγιση. Πιθανώς χρειαζόμαστε κάποιες συνεδριάσεις ακόμα για να πείσουμε και τους συναδέλφους αλλά αν θέλουμε να επιτύχουμε πράγματα πρέπει να διευρύνουμε την βάση μας. Γι' αυτό ακριβώς είναι σωστά τα ολοκληρωμένα αυτά έργα. Αυτό το οποίο είπε Χέλγα για το ΦΠΑ και τη συγχρηματοδότηση και όλα αυτά και με αυτά συμφωνώ ανεξαρτήτως του ότι και στον κανονικό κανονισμό του ε, προϋπολογισμού ούτως ή άλλως το έχουμε ψηφίσει αυτό ήδη. Δηλαδή επιλέξιμος ο ΦΠΑ εκεί όπου οι ε, ΜΚΟ δεν είναι σε θέση ε, να χρηματοδοτηθούν από εθνικούς προϋπολογισμούς. Και δήμοι η περιφέρειες δεν πληρώνουν ΦΠΑ ούτως ή άλλως, οπότε δεν τίθεται ζήτημα και με τα λίγα λεφτά που έχουμε πρέπει λεφτά που έχουμε για το live να τα χρησιμοποιούμε σωστά. Πετυχαίνουν πολλά αλλά σε σχέση με τους εθνικούς προϋπολογισμούς είναι λίγα και πρέπει με τα λίγα λεφτά που έχουμε να γεμίσουμε, δεν ξέρω, και τα α, των, τα εθνικά ταμεία να πληρώνουμε και ΦΠΑ από πάνω 20%. Δεν νομίζω. Οπότε συμφωνώ με την Χέλγα και παρακαλώ τους συναδέλφους να α, ακολουθήσουν την δική της ε, τακτική. Ευχαριστώ, Σαλβαδόρ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εγώ δεν έχω καμία αντίρρηση σε αυτά τα οποία μας λέει η Χέλγα και σε αυτά που προσθέτει η Γιούτα. Απλώς επιστήνω την προσοχή σας στην τροπολογία 5 και στην 6 της έκθεσης της Helga Τρούπερ όπου γίνεται μία σαφής αναφορά στα ποσοστά του Γενικού Προϋπολογισμού της Ένωσης. Εμείς σκεφτήκαμε στη ΣΟΥΡΕ, στην Επιτροπή ΣΟΥΡΕ, ότι για το 2014 δεν θα έπρεπε να εντάξουμε μέσα στα πλαίσια της ε, δημοσιονομικής συζήτησης ε, συζητήσεις ε, για το, το συνολικό μέγεθος του για το πώς σχηματίζεται συνολικά ο προϋπολογισμός έπρεπε να έχουμε το συνολικό μέγεθος Μήπως θα μπορούσαμε λοιπόν να εξηγήσουμε αυτήν την αντίφαση μεταξύ των ποσοστών που ε, συμπεριλαμβάνονται εδώ με την γενική συμβατότητα που διατηρήσαμε όταν συντάξαμε την έκθεση ΣΟΥΡΕ. Εγώ δεν έχω κατά τα άλλα καμία αντίρρηση ουσίας στο σχέδιο έκθεσης. Πολύ ωραία. Η Χέλγα. Ευχαριστώ τους συναδελφούς για τις συνεισφορές τους. Ευχαριστώ ειδικά τη Γιούτα που υποστηρίζει την προσέγγισή μου. Υπάρχει ένα πολιτικό επιχείρημα. Το αν θα πρέπει να αναφέρουμε τα ποσοστά. Κάναμε μια γενική συζήτηση, αλλά αποφάσισα να μην βάλω νούμερα. Δεν πρέπει να το κάνουμε αυτό αυτή τη χρονική στιγμή. Θα πρέπει να πούμε πολιτικά τι θέλουμε να πετύχουμε με το live και γιατί θα πρέπει να είμαστε πιο φιλόδοξοι σε σχέση με τις δηλώσεις μας που έχουμε κάνει απέναντι στην κλιματική πρόκληση, στην προστασία του περιβάλλοντος, την προστασία της βιοπικιλότητας. Γι' αυτό αποφάσισα να μην βάλω νούμερα. Νομίζω ότι είναι καλύτερο, είναι πιο ενδεδειγμένο και συνάδει με τους κανόνες και τις αποφάσεις μας. Φυσικά θα πρέπει να δούμε τελικά πώς θα προχωρήσουμε. Πιστεύω ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Ούτω ή άλλω και σε άλλου τομεί το κάναμε. Με το πρόγραμμα για τη διαβίου μάθηση. Δεν νομίζω ότι καταστρέφει το πλαίσιό μας. Είναι μια σαφής πολιτική δέσμευση για αυτό που θέλουμε να υπάρξει, αυτό που θέλουμε να επιτύχουμε. Ευχαριστώ. Υπάρχει ευρεία συνένεση. Όλοι θέλουν να υποστηρίξουν αυτό το πρόγραμμα. Στην πρώτη μου θητεία στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είμαι εισηγητή του προπολογισμού και ήμουν ο πατέρα, ο εφευρέτη του, του LIFE. Βρήκα και τη λέξη και το περιεχόμενο. Δηλαδή, δημοσιονομικό μέσο για το περιβάλλον. Στα αγγλικά φτιάχνει έτσι ένα ωραίο ήχο. Τότε δεν τα καταφέραμε, αλλά ίσως η Χέλγα τα καταφέρει. Αυτό που θέλαμε ήταν να φτιάξουμε ένα διαφορετικό ταμείο. Αυτή είναι η ιδέα τότε. Ε, υπάρχουν οι πολιτικέ διαφορετικέ, υπάρχει η κοινωνική πολιτική, πολιτικέ συνοχή κτλ. και η προστασία του περιβάλλοντο. Ε, τότε τη λέγαμε βιώσιμη ανάπτυξη. Μάλλον τώρα τη λέμε βιώσιμη ανάπτυξη. Όλοι θέλουμε αύξηση των πόρων, αύξηση των μέσων. Θα το βάλουμε στην ομοδότηση. υπό τη μορφή προτείνει η Χέλγκα. Όπως λέει ο Σαρβατόρ, υπάρχει πρόβλημα αρχής σε σχέση με τη θέση που υιοθετήσαμε με το contact group, με την ομάδα επαφής. Θα πρέπει να δούμε τι σκέφτονται οι δύο Θα δούμε τις τροπολογίες και ανάλογα θα αποφασίσουμε. Θυμίζω το χρονοδιάγραμμα. Προθεσμία για τις τροπολογίες αύριο. Πολύ γρήγορα. Ναι, ναι, εντάξει. Θα περάσετε τη νύχτα φτιάχνοντας, συντάσσοντας τροπολογίες. 6 Σεπτεμβρίου η έγκριση και θα ψηφίσουμε 19 Σεπτεμβρίου στην Επιτροπή Περιβάλλοντος και αυτό θα επιτρέψει στην Επιτροπή Περιβάλλοντος να διαπραγματευτεί με το Συμβούλιο εμπρόθεσμα. Ευχαριστώ την Έλγα. Ήρθε η ώρα 19. Το 19. Α, μου είπατε ότι ήθελε να το αναβάλει. 19. Ήθελε να σας κάνει να μιλήσετε νωρίτερα. Λοιπόν, καινοτόμα, καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα στο πλαίσιο της, του επομένου πολιετούς δημοσιονομικού πλαισίου. Ναι, εγώ προσπάθησα να το προλάβω, να, να το βάλω λίγο νωρίτερα το κείμενο, γιατί πάντα όταν μιλάμε για PDP, πάντα πέμπτη απόγευμα είναι. Λοιπόν, όπως λέει αυτή η έκθεση για τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά σχέδια και για το νέο PVP 2014-2012, η έκθεση θα είναι πολύ γενική. Δεν θα μπούμε στις λεπτομέρειες του κάθε δημοσιονομικού μέσου. Δεν ήταν στόχος ούτε της έκθεσης, ούτε αυτής της Επιτροπής. Στο πρώτο τμήμα της έκθεσης αυτό που προσπαθήσαμε είναι να δώσουμε μία πιο, όσο το δυνατόν πιο απλή εξήγηση για το ποια είναι τα δημοσιονομικά μέσα, γιατί χρησιμοποιούνται και σε τι χρειάζονται. Και ο στόχος αυτών των μέσων είναι να, να δώσουν κίνητρα, επενδυτικά κίνητρα στην κοινωνία. Παίζουν ένα καταλητικό ρόλο Δηλαδή μπορούμε έτσι να κινητοποιήσουμε περισσότερους πόρους και να χρηματοδοτήσουμε τα στρατηγικά σχέδια για την ανάπτυξη της Ένωσης που με άλλο τρόπο δεν θα μπορούσαμε να καταφέρουμε. Διότι αυτά τα χρηματικά, χρηματοδοτικά μέσα λειτουργούν όταν υπάρχει πρόβλημα στην αγορά και Έχουμε το κεφάλαιο κινδύνου, επενδυτικό κεφάλαιο, μετά έχουμε τα μέσα χρέους που χρησιμοποιούμε ως εγγύηση, αντεγγύηση. Έχουμε την κατανομή ε, του ρίσκου με αντιπαροχές. Λοιπόν, το ρίσκο, κίνδυνος που συνεπάγεται η χρήση των δημοσιονομικών μέσων για τον προϋπολογισμό. Εγώ λέω ότι ο κίνδυνος είναι πάρα πολύ περιορισμένος και ελεγμένος, διότι στη χειρότερη περίπτωση θα μπορούσαμε να χάσουμε μόνο το ποσό το οποίο δεσμεύσαμε στη γραμμή του προϋπολογισμού, το ίδιο, τον ίδιο κίνδυνο δηλαδή με μία επιδότηση που είναι χαμένο χρήμα μετά δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιδοτήσεις αλλά ούτε και ως ε, πρόσχημα για να μειώσουμε τον προϋπολογισμό. Στην άλλη, στο άλλο τμήμα της έκθεσης προσπαθώ να αναλύσω την πρόταση της Κομισιόν ε, υποβάλλοντας προτάσεις ή αιτήματα. Ε, την πρόταση της Κομισιόν θεωρούμε ότι πάει προς την σωστή κατεύθυνση και μειώνουμε τα χρηματοδοτικά μέσα και επικεντρώνουμε καλύτερα τη δράση αυτών των μέσων. Θεωρούμε ότι είναι πολύ καλή ιδέα να δημιουργηθούν πλατφόρμες κεφαλαίου χρέους. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε απλούστευση και μεγαλύτερη συνοχή. Και πρόκειται για κάτι το για το οποίο υπήρξε πολλή ζήτηση. Άλλη ιδέα της ε, Κομισιόν είναι να συνδυάσουμε στην πολιτική ε, συνοχή ε, ε, δάνεια και επιδοτήσεις. Ένα, ένα 600 δις. Ε, εμείς ε, πρέπει να κινητοποιήσουμε το απαραίτητο κεφάλαιο αν θέλουμε να προχωρήσουμε. Λοιπόν, εμείς πρέπει να εξηγήσουμε ότι για να γίνει κάτι τέτοιο πρέπει να έχουμε ένα διαφανές νομικό πλαίσιο, σαφείς κανόνες και σαφήνια στα χρηματοδοτικά μέσα και οι επανεισρωές, τα reflows θα πρέπει και αυτά να χρησιμοποιούνται. Και καταφέραμε εμείς να κάνουμε ένα βήμα με το Συμβούλιο και θα χρησιμοποιήσουμε μέγα μέρος των reflows. Και μετά έχουμε και τις αξιολογήσεις, τις, ε, τους ελέγχους εξάντε, διότι εμείς βρισκόμαστε σε μια κατάσταση όπου τα χρηματοδοτικά μέσα πρέπει να παρεμβαίνουν και βρισκόμαστε σε μία κατάσταση ε, επιδοτήσεων μέσα σε ένα σύστημα αγοράς. Εμείς πρέπει να δούμε πώς λειτουργούν όλα αυτά τα μέσα. Πρέπει να, να τα τροποποιήσουμε και να τα αξιολογήσουμε. Θα ζητήσουμε λοιπόν για την αξιολόγηση μία ετήσια έκθεση όπου θα έχουμε τύπους ε, κονδυλίου, θε, θεματικές, ε, κράτος μέλος για να έχουμε όλες τις πληροφορίες. Ζητούμε επίσης ευελιξία. Πολύ χρησιμοποιούμε αυτόν τον όρο ευελιξία στον προπολογισμό και χρειάζεται και για, τη χρημα... για τα χρηματοδοτικά μέσα. Εν ώψη του 2020 ξέρουμε πώς λειτουργούν οι χρηματοπιστωτικές αγορές. Ποια είναι και η κοινότητά τους, αλλά δεν και δεν ξέρουμε και πώς θα χρησιμοποιήσουν τα μέσα που θα έχουμε στη διάθεσή μας. Μπορεί να έχουν κουσούρια άλλα μπορεί να χρειάζονται περισσότερο χρήμα και άλλα λιγότερο. Οπότε η αρχή του προπολογισμού πρέπει να είναι αυτή η οποία ετησίως θα αποφασίζει τα ποσά τα οποία θα αναδώσουμε, με τα οποία θα πρικοδοτήσουμε το κάθε χρήμα. Ε, χρήμα ε, το πιστοτικό μέσο. Πρέπει λοιπόν να έχουν ένα θετικό αποτέλεσμα στην ευρωπαϊκή οικονομία αλλά είναι όμως περιορισμένα ως προς τα σχέδια, ως προς τις επενδύσεις μέσω και βραχυπρόθεσμα και υπάρχει και ένα άλλο βήμα που πρέπει να κάνουμε. Εμείς ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ αποταμίευση, ιδιωτική αποταμίευση, που ψάχνει ασφαλή με, ε, ε, ε, ασφαλείς επενδύσεις. Θα πρέπει λοιπόν εμείς να κοιτάξουμε να θέλξουμε αυτό το κεφάλαιο για να χρηματοδοτήσουμε τα σχέδια του 2020. Πρέπει λοιπόν να βρούμε ένα νέο ε, χρηματοπιστωτικό μέσο που θα μπορέσει να ε, συνδυάσει και τις ανάγκες Ευρωπαϊκής Ένωσης μακροπρόθεσμα για διάφορα σχέδια αλλά και να τραβήξει αυτό το ιδιωτικό κεφάλαιο. Ζητούμε λοιπόν κάτι παραπάνω για να μπορέσουμε να είμαστε από την Κομισιόν για να είμαστε πιο φιλόδοξοι στα σχέδιά μας. Περιμένω τα, σχέδια, τα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ, Έιντερ. Ο Ντομινίκ Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είμαι σκιώδης εισηγητής του ΕΛΚΑ. Γι' αυτό κοίταξα προσεκτικά την έκθεση. Συνήθως ε, συγχαίρουμε τον εισηγητή, την εισηγητή για τη δουλειά της. Αλλά εδώ το αξίζει κιόλα. Γιατί την έχει προβληματίσει πολύ ενδελεχώς ε, το θέμα και η δουλειά της είναι πολύ καλής ποιότητας. Είναι, δεν είναι τόσο εύκολο με ένα τόσο πυκνό κείμενο. Θα υποστηρίξουμε βέβαια το σχέδιο έκθεσης όπως παρουσιάζεται και υπό τη μορφή που παρουσιάζεται και στην ουσία του το ευστηρίζουμε. Θέλουμε και εμείς να βάλουμε το λιθαράκι μας στο οικοδόμημα όμως. Υπάρχουν κάποια στοιχεία που μας ενδιαφέρουν πιο πολύ και πρέπει να τονιστούν λίγο περισσότερο. Καταρχάς, για την ευρωπαϊκή προστιθέμενη αξία. Δηλαδή, τι εξυπηρετούν αυτά τα μέσα. Δεύτερον, υπόθηκε, αλλά καλό θα ήταν να το πούμε πιο λεπτομερώς. Διάφορες περιπτώσεις επενδύσεων και να τονίσουμε ότι όλα αυτά ε, διέπονται από τον δημοσιονομικό κανονισμό, έτσι, τέλος πάντων τον νέο δημοσιονομικό κανονισμό. Ούτως ώστε Ξέρουμε βέβαια ότι κάθε φορά το Συμβούλιο ε, βάζει παρατήματα και τα σερβίρει όλα αυτά μέσα σε μια γενική σάλτσα προσθέτει πράγματα που δεν είναι επιθυμητά κάθε φορά. Τέλο πάντων, η συζήτηση γίνεται στα πλαίσια του δημοσιονομικού κανονισμού. Θα πρέπει να πούμε λοιπόν εμεί ξεκάθαρα τι θέλουμε σε αυτή την περίπτωση. Να τονίσουμε επίση την ευθύνη τη Ένωση και την ορατότητα που θα πρέπει να έχει η παρέμβαση τη Ένωση. Γιατί όσο πιο περίπλοκο είναι το προϊόν, ε, τόσο πιο πολύ εξαφανίζεται η Ευρώπη μέσω σε αυτού του ενδιάμεσου μηχανισμού. Ε, ε, πίσω από τους υπεύθυνου για τα προγράμματα. Εμείς θα πρέπει να θέλουμε αυτή η ορατότητα, η διαφήμιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να μην εξαφανιστεί ε, σε αυτά τα καινοτόμα χρηματοπιστωτικά μέσα. Τελειώνοντας, να πω το εξής. Το είπε καλά η κυρία Γκάρδια Ταβάλ. Υπάρχουν εκατομμύρια, για να μην πω δισεκατομμύρια, στις χρηματαγορές που είναι στα χέρια συνταξιοδικών ταμείων, ασφαλιστικών ταμείων, οι equity funds που ψάχνουν προγράμματα σταθερά, εγγυημένα και μη κερδοσκοπικά. Λοιπόν, αν η Ευρώπη έχει καλά έργα, καλά προγράμματα και μπορεί να εγγυηθεί και ένα τμήμα τους, τότε τη στιγμή που έχουμε πρόβλημα τα, ε, πόρων και κρατικών κονδυλίων, έτσι, εκείνη τη στιγμή Μπορεί να υπάρχει μια σύγκληση ανάμεσα στην αποταμίευση της, των ιδιωτών και το χρήμα αυτό να πάει εκεί πέρα και να γονιμοποιήσει αυτά τα φυτόρια. Κάτι που θέλω να προσθέσω στην έκθεση. Η φαντασία των χρηματιστών είναι χωρίς όρια αν βάλουμε στην αγορά προϊόντα χρηματοπιστωτικά υπό την ε, μορφή των νέων χρηματοπιστωτικών μέσων και τα προϊόντα αυτά είναι ελκυστικά, φτάσουν σε μια κρίσιμη μάζα, σε έναν όγκο και μας εξασφαλίσουν και ασφάλεια αλλά και ρευστότητα, τότε μπορούμε να φανταστούμε ότι αυτά τα προϊόντα θα τυπλοποιούνται, θα είναι περίπλοκα ή θα χρησιμοποιούνται σε συνθήκες που δεν θα είναι πολύ αποδοτικές. Ε, δεν αποκλείεται. Ειδικά όταν είναι επιτυχημένα μερικά, αυτό συμβαίνει. Και νομίζω ότι θα ήταν σημαντικό να είμαστε προσεκτικοί, ούτω ώστε αυτή η περιπλοκότητα των μέσων, η αγορά τα κάνει περίπλοκα, ε, να μην οδηγήσει στην, στη χρήση τους με τρόπους που δεν, μας, που δεν είναι αποδοτικοί για μας. Όσο δεν είμαστε προσεκτικοί για το θέμα, αυτό θα συμβαίνει. Ε, επίσης, η Ένωση προς το παρόν δεν έχει πιστέψει στην επιτυχία αυτού του μηχανισμού. Αν λειτουργήσει όμως επιτυχώς, μπορούμε να έχουμε προβλήματα εν συνεχεία με αυτά τα προϊόντα. Εκεί θα πρέπει να προσέξουμε ακόμα περισσότερο. Η ευρωπαϊκή εγγύηση είναι περιορισμένη, το ξέρουμε. Και το είπε και η συγκήτρια. Η δέσμευση της Ένωσης σε δημοσιονομικό πλαίσιο περιορίζεται στο ποσό που εγκρίνει η Δημοσιονομική Αρχή. Αλλά δεν είναι μόνο το χρήμα σε αυτήν την ιστορία και σε αυτό θέλω να τονίσω. Σε αυτό θέλω να σταθώ. Οι χρηματαγορές έδειξαν μια πραγματογνωμοσύνη στα πιο διαφορετικά προϊόντα. Δεν μπορούμε να είμαστε σίγουροι λοιπόν ότι όλα αυτά θα γίνουν ε, με άμεμπτο τρόπο. Ευχαριστώ Ντομινίκ. Πιστεύω όπως το είπαν η Σιγήτρια και το Ντομινίκρη και αυτό το θέμα είναι ουσιαστικό. Χρειαζόμαστε να δημιουργήσουμε ή να ενισχύσουμε μέσα για να αντιμετωπίσουμε μια κατάσταση που είναι πάρα πολύ ιδιόμορφη και περίεργη όπου έχουμε πάρα πολύ χρήμα τεράστιες ποσότητες έχουμε τα εθνικά, εθνικά ταμεία κρατικά ταμεία, ε, έχουμε τα ισοζύγια πληρωμών με τα πλεονάσματα τους των αναδειωμένων χωρών και των ε, ε, χωρών παραγωγών πετρελαίου. Έχουμε επίσης και όλοι αυτοί, αυτά, αυτές τις χρηματοπιστωτικές μάζες που έχουν συσσωρευτεί αυτά τα τελευταία χρόνια. Εγώ έφαγα τις προάλλες με τον Jean-Claude που έλεγε ότι στα 10 χρόνια η μάζα χρημάτων που πλανάται επί των κεφαλών μας και που μπορεί κάποια στιγμή να πέσει πάνω σε μια συγκεκριμένη επένδυση, μια χώρα ή οτιδήποτε άλλο, έχει πολλαπλασιαστεί επί 35. Υπάρχει πραγματικό χρήμα, ψεύτικο χρήμα, κερδοσκοπία ή μη κερδοσκοπία, όλα αυτά είναι πολύ μπερδεμένα. Αλλά υπάρχει μία μάζα χρήματος έτοιμη να επενδύει και να έρθει να, να, ε, και να επενδύσει, φτάνει να έχει ασφάλεια και απόδοση. Και με, έχουμε την, με, την, αυτή την... Ε, ε, ε, αλλαγή, τη μεταρρύθμιση. Δηλαδή ένα μία βραχυπρόθεσμη κατάθεση να την μετατρέπουν σε μακροπρόθεσμες ε, καταθέσεις ή επενδύσεις. Τώρα οι τράπεζες σήμερα μειώνουν, ε, βλέπουν μέσα από την κρίση να μειώνονται αυτές τους οι δυνατότητες και λόγω της ευπάθειας αυτών που έκαναν τις κερδοσκοπικές επενδύσεις αλλά έχουμε και τους κανόνες ε, Βασιλεία 3, Solvency 2, Omnibus ε, δεν ξέρω ποιον αριθμό που τους επιτρέπουν να αυξάνουν το κεφάλαιό τους, ε, να αυξη... το, το, το, παθητικό και ενεργητικό και δεν τους επιτρέπουν να επενδύουν τάντο. Λοιπόν, αποτέλεσμα όλης αυτής της ιστορίας. Έχουμε το πρόβλημα, το, το σχέδιο των χρηματοδοτικών μέσων, καινοτόμων χρηματοδοτικών μέσων που, μιλήσαμε, που μιλάμε τώρα και πολύ πιθανόν, όπως λέει και ο Ντομινίκ Ρικέ, πολύ σύντομα να μας προτείνουν για να μπορέσουμε να έχουμε και μια κριτική μάζα και να έχουμε μεγαλύτερη ορατότητα, μικρότερα επικότητα, να έχουμε μεγαλύτερη ρευστότητα στην αγορά, να τα ε, ενώσουμε όλα αυτά και να έχουμε ένα φάκελο σχεδίων. δηλαδή ή με τις ομολογίες, με, με τις μετοχές, ε, φακέλους μετοχών και τα λοιπά ε, και καινοτόμων σχεδίων. Είδαμε όμως με τις μετοχές τι γίνεται. Ε, ευχαριστώ τον την εισηγήτρια και τους ομιλητές διάγραμμα για αυτήν την έκθεση 19 Ιουλίου, η προθεσμία για τις τροπολογίες έγκριση 6 Σεπτεμβρίου. ...6 Σεπτεμβρίου θα έχουμε ένα σωρό ψυχοφορίες. Σημείο 8. Αλία. Αλλάζουμε θέμα. τελευταίο απόγευμα πριν από τις διακοπές, οπότε διαφοροποιούμε την ψυχαγωγία μας. Ο συνάδελφος Αλφόνση ήδη ψαρεύει στα νυχτά της Κορσικής, αλλά η Ζαμπέλη είναι ακόμη εδώ και τον αντικό του στοθεί. Αλία της Βόρειας Θάλασσας κατά της Αλίας στην Κορσική. Εγώ αντικαθιστώ εδώ τον Φρανσουά Αλφόνση, για να σας παρουσιάσω την υποστήριξη σε αυτό το σχέδιο, η Κομισιόν διαπραγματεύτηκε αυτό το νέο πρωτόκολλο αλίας με την Δανέζικη κυβέρνηση για τη Γρυλανδία. Στην από την 1η Ιανουαρίου του 2013 έχουμε αντιπαροχές της τάξης των 17 δισεκατομμυρίων και, και διαφόρων εκατομμυρίων το χρόνο. Έχουμε ένα ετήσιο ποσό 15 εκατομμύρια ευρώ για την πρόσβαση στην αποκλειστική ζώνη αλλίας της Γρυλανδίας ε, για ένα ποσό 2.503.000 και κάτι ψηλά για να υποστηρίξουμε την πολιτική αλίας της Γρυλανδίας. Επίσης ε, προβλέπονται και διάφορες διατάξεις για την αηφορία της αλίας στις ε, ακτές της Γρυλανδίας με ποσοστό στις αλίας και βοηθητικά μέτρα, επιστημονική συνεργασία, ε, εφαρμοστικές ε, λεπτομέρειες που πρέπει να καλύπτουν, ζητουμένων που πρέπει να καλύπτονται από τα πλοία και τα λοιπά, τα ευρωπαϊκά πλοία. Υποστηρίζει την έκθεση και θα σας στείλει από την Κορσική εντός των ημερών την έκθεσή του. Ωραία. Η στο Παρτίδο Ποπουλάρ. Αυτή η λαρότητα της δεξιάς, εκτός από αυτήν, έχουμε να πούμε τίποτα άλλο, να κάνουμε άλλες παρατηρήσεις. Ευχαριστώ για αυτή την έκθεση. Θα στείλουμε στη μετάφραση την έκθεση στις 20 Ιουλίου. Δεν έχουμε καταληκτική ημερομηνία για τις τροπολογίες, πρέπει να βάλουμε μία. Και η ψηφοφορία θα γίνει πού, πότε. Α, στην Επιτροπή Προπολογισμού στις 6. Ούτως ώστε να είναι έτοιμη για την Επιτροπή Αλίας που ψηφίζει τον Οκτώβρη. Θα πρέπει να πούμε στους συναδέλφους και ποια είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες, έτσι. Ευχαριστώ, Φρανσουά Αλφόνση, που ήσασταν τόσο σύντομο στην παρουσίαση, δηλαδή, εκπρόσωπος. Είναι μια διαδικασία σύμφωνη γνώμη. Λέμε δηλαδή α, ναι ή όχι. Δεν υπάρχουν τροπολογίε, άρα δεν υπάρχει και προθεσμία. Θα ψηφίσουμε ναι την επόμενη φορά λοιπόν, έτσι. Πραγματική δημοκρατική διαδικασία, κορσική μέθοδος, να Μόνικα καλό στη Μόνικα σούπερσταρ με τρεις εκθέσεις που συμπληρώνουν την ε, έκθεση του Ντομικίν Ρικέ για το Ταμείο Ιστορικής Ασφάλειας. Προτείνω στη Μόνικα να μας παρουσιάσει και τις τρεις εκθέσεις μαζί. Αγαπητέ κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, σας ευχαριστώ για το ότι μπορώ να παρουσιάσω και τις τρεις αυτές μαζί είναι οι γνωμοδοτήσεις της Επιτροπής μας για το Ταμείο Ασύλου, Εσωτερικών Συνόρων και Βίζας, αλλά και τις γενικές διοικητικές διατάξεις για τα δύο αυτά ταμεία ασύλου και μετανάστευση και εσωτερικής ασφαλής. Από όσο ξέραμε υπήρχαν μέχρι πρόσφατα τέσσερα ταμεία, ταμείο ενσωμάτωσης προσφύγων, επαναπροώθησης και μετανάστευσης και το, πρόγραμμα, και τα δύο προγράμματα αυτά και διαφορετικοί κανόνες διοίκησης για το κάθε ένα. Η πρόταση της Κομισιόν για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο προβλέπει προσεχώς δύο μόνο ταμεία και κυρίως ενιαίους κανόνες διοίκησης. Είναι μια καλή ε, πρόταση αυτή και νομίζω πως ε, συμφωνεί και με αυτά τα οποία ε, θέλει και το Κοινοβούλιο. Θα πρέπει να υπάρχει ε, μια ε, χωριστή διαχείριση των μέσων και με ένας διάλογος πολιτικής με τα κράτη-μέλη για να ορίζονται από κοινού οι στόχοι της πολιτικής, όπως ήδη σήμερα συμβαίνει στην ε, διαρθρωτική πολιτική. Θα υπάρχει επίσης μια κεντρική διαχείριση των κοντιλίων για τα λεγόμενα μέτρα της Ένωσης, για τα μέτρα ανάγκης, για τα δίκτυα και την ανάπτυξη νέων πληροφοριακών συστημάτων υπό τον τίτλο «Έξυπνα σύνορα». Κατόπιν έχουμε μια πολυετή, ένα πολυετή προγραμματισμό. Σε κάποια προγράμματα είχαμε ετήσιο μόνο προγραμματισμό και βεβαίως αυτό δημιουργεί πολλά προβλήματα όσον αφορά την αποδοχή τους. Θα έχουμε λοιπόν σταθερά αλλά και μεταβλητά ποσά. Θα έχουμε ένα 75% που θα είναι ο κανονικός ε, ρυθμός, το ε, κανονικό ποσοστό χρηματοδότηση χρηματοδότησης σε 90% σε κάποιε περιπτώσει και σε στρατηγικά έργα θα φτάσει στο 100%. Επίσης είδα προσεκτικά όλα τα νούμερα και ε, ξεπλάγει από το ότι κάποια από αυτά δεν έχουν επαρκή ποσά και πραγματικά αναμένω πώς θα χρηματοδοτηθούν αυτά. Αν δούμε παραδείγματος χάρη το νέο κέντρο κυβερνοεγκλήματος. Πώς θα γίνει κάτι τέτοιο αν ταυτόχρονα η Europol παίρνει μείον 10% χρηματοδότηση. Πού θα βρει προσωπικό. Δεν ξέρω, μου φαίνεται κάπως περίεργο και σε άλλα σημεία του υπερπολογισμού υπάρχουν ερωτήσει. Οπότε η πρόταση αυτή, η πολιετής, ε, παραμένει νομίζω κάτω και από την πρόταση του 2013. Οπότε θα πρέπει να συζητήσουμε για το θέμα ασύλου, μετανάστευσης, συνόρων. Αναμένουμε πάρα πολλές ε, ερωτήσεις και βεβαίως ε, θα πρέπει να ε, αναμένει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο κάποια απάντηση τώρα για την διάρθρωση των ταμείων, η αναδιάρθρωση της εσωτερικής διοίκησης κατά την άποψή μου είναι κάτι το επιτυχημένο με τους ενιαίους αυτούς ε, κανόνες. Ε, τώρα μας απασχολεί το τι πρέπει να κάνει η Κομισιόν με τις ε, πράξεις κατεξιοδότηση καθώς καμιά φορά η εκτροπή Προπολογισμού χάνει την εικόνα και την εποπτεία τι συμβαίνει, τι δεν συμβαίνει Οπότε θα πρέπει να περιοριστούν οι πράξη κατεξιοδότηση μόνο στα της εκτέλεσης σε συγκεκριμένα πράγματα, αλλά όχι την πολιτική ε, διαμόρφωση ε, της ε, πολιτικής που θα ακολουθούν βεβαίως αυτές οι υπηρεσίες και υπάρχει και το θέμα της διαφάνειας των κονδυλίων και θα πρέπει να υπάρχει οπωσδήποτε και μια ξεκάθαρη ευρωπαϊκή προσθεμένη αξία. Οι ειδικέ μου τροπολογίες ε, πηγαίνουν στο ότι πρέπει εκεί όπου έχει διαπιστωθεί διοικητική αδυναμία των κρατών μελών να ενισχυθούν από την Κομισιόν. Αυτό βεβαίως δεν απαλλά τα κράτη-μέλη από την ευθύνη τους, αλλά ε, βεβαίως όταν κάτι δεν ε, λειτουργεί θα πρέπει από κοινού να προσπαθήσουμε να βελτιώσουμε την διοικητική ικανότητα στα κράτη-μέλη αυτά. Επίσης, ε, λογικό, λογική είναι η ε, ευνηδιαστική επιτοπή έλεγχη, επίσης η χρηματοδότηση κάποιων μέτρων κατά 100 της 100 ε, ε, πλην των περιπτώσεων βεβαίω όπου έχουμε εθνικό προσωπικό δεν μπορούμε να το πληρώνουμε από κονδύλια της ε, Ένωσης. Ε, επίσης θα πρέπει να δούμε στον πολιτικό διάλογο και την συμμετοχή των υπηρεσιών αυτών για να μπορέσουν να πούν την άποψη της υπηρεσίας τους και να μην εκπροσωπούνται μόνο μέσω της Κομισιόν. Να έχουν και αυτή λόγο στις ε, συζητήσεις αυτές. Το κείμενο συμφωνεί με τον ε, νέο δημοσιονομικό κανονισμό και τους ε, βελτιωμένους κανόνες για την διαχείριση κονδυλίων. Εν τω μεταξύ δεν χρειαζόμαστε μία μόνο προχρηματοδότηση, αλλά ετήσια προχρηματοδότηση για να υπάρχει συνέχεια, γιατί υπήρχαν μέχρι τώρα προβλήματα, προβλέπονται 3,52 δις 31% ε, για τα εθνικά προγράμματα ε, μεταξύ των οποίων και της Λιθουανίας 31% ε, για τα έξυπνα σύνορα και βεβαίως έχουμε και το Ταμείο για τα εξωτερικά σύνορα και τις θεωρήσεις και θα πρέπει να δούμε και την προσθέμενη αξία σε σχέση με τις ε, τρίτες χώρες και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να κινηθούν στο πλαίσιο των ε, στόχων που έχουμε θέσει για να μην υπάρχουν άλλοι επικαλύψεις και επαναλήψεις ε, πραγμάτων που γίνονται σε εθνικό επίπεδο όσον αφορά το Ταμείο Ασύλου και Μετανάστευσης έχουμε ένα 80% που θα προγράμματα, 20% κεντρική διαχείριση. Οι τροπολογίε μου εδώ πέρα είναι οι τυποποιημένε, δηλαδή λογοδοσία, διαφάνεια, συμπληρωματικότητα όπως συναποφάσισαν και οι συντονιστές και βεβαίως και σε αυτό τον κανονισμό πρέπει να δούμε την, τον αριθμό των πράξεων κατεξοδότηση που είναι αρκετές. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε παρατηρήσεις. Πριν τελειώσουμε με τα χρηματοπιστωτικά μέσα, είναι κάτι που έπρεπε να πω πριν. Γιατί βλέπω τους αδέλφους να φεύγουν με λαφρά πηδηματάκια. Χθες το βράδυ ε, δείπνησα, όλα για δείπνα σας λέω, με την Κόνι ε, Χέντγκαρτ, πολύ γοητευτική κυρία, υπεύθυνη για την πολιτική περιβάλλοντος και τη σχέση μεταξύ περιβάλλοντο και ενέργεια. Και νόμιζα ότι κατάλαβα από την παρουσίαση που έκανε ότι από 1η Ιανουαρίου του 2013 θα εφαρμοστεί το σύστημα πώληση σε δημοπρασία των δικαιωμάτων εκπομπής αέριων του θερμοκηπίου, το ETS. Ένα σύστημα που θα ισχύει. Η αγορά του ETS λειτουργεί με δωρεάν εκπομπές, για να το πω έτσι, και συνεχεία πληρώνουμε στη δευτερογενή αγορά από το 2005. Και από την 1η Ιανουαρίου 2012, καλύτερο ο πρόεδρος, συνήθως κανονικά οι αεροπορικές εταιρείες πρέπει να πληρώσουν. Ξέρετε ότι υπάρχει μια διένεξη με τις εταιρείες που εξυπηρετούν την Ευρώπη, αλλά που δεν έχουν τη βάση τους στην Ευρώπη. Και από την 1η Ιανουαρίου 2013 όλες οι ρηπογόνες δραστηριότητες πρέπει να πληρώνουν οι υπεύθυνοι για αυτές. Η ιδέα της ε, Επιτρόπου Χέντγκαρτ ήταν να πληρωνουν υπευθυνοι για ένα τμήμα αυτών των πόρων που θα προκύψουν από αυτή την πώληση δικαιωμάτων για ρήπους για να χρηματοδοτήσουμε κάποιες πολιτικές για το περιβάλλον. Η ιδέα είναι πολύ ενδιαφέρουσα αυτή καθεαυτή. Εγώ όμως διερωτώ μου κάτι που δεν, δεν τη ρώτησα την ίδια, αλλά το λέω στη γραμματεία, στους συναδέλφους των αυτών που ασχολούνται με τα χρηματοπιστωτικά και με τους ίδιου πόρου. Έθεσα λοιπόν το εξή ερώτημα. Και η Επίτροπη λοιπόν το έχει θέσει και επίσημα νωρίτερα. Τώρα, αν το θέτει, το καλύτερο έστω και τώρα. Ποιο είναι ο δικαιούχο αυτών των πόρων, ποιο είναι αυτό ο προπολογισμό, δηλαδή ποιο είναι αυτό το κονδύλι, για εκείνο είναι ευρωπαϊκό σύστημα, θα έπρεπε κανονικά να, πάει αυτό το, να πάνε όλα αυτά τα χρήματα στο ενωσιακό προπολογισμό. Αλλά μέχρι στιγμή, έτσι όπω είναι διατυπωμένο ο κανονισμό για το σύστημα ανταλλαγή εμπορία ε, των εκπομπών, πάνε στου εθνικού ε, προπολογισμού. Αν μπορέσουμε να πάρουμε ένα τμήμα από αυτού του πόρου, θα πρέπει να χρηματοδοτήσει ένα χρηματοδοτικό μέσο ad hoc, θα θεωρηθούν ήδη πόροι, ένας επιπλέον ίδιος πόρος καινούριο. Πριν από λίγους μήνες, όταν προσπαθήσαμε να κάνουμε ένα κατάλογο με τους πιθανούς καινούριου νέους πόρους που θα τροφοδοτήσουν τον ενωσιακό προϋπολογισμό, κάτι είχαμε ψελίσει για αυτό το θέμα. Αλλά τότε ο Λεβαντόφσκι και άλλοι επίτροποι μας είχαν πει, όχι, έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Δεν πρέπει να ξανανοίξουμε αυτή την ιστορία, αποκλείεται, αλλά αν η Επιτροπή αλλάζει γνώμη ή ακούγονται νέε φωνέ στην Κομισιόν, ίσως θα πρέπει να το ξαναδούμε αυτό το πράγμα. Ε, Μόνικα ε, pour Ευχαριστώ Μόνικα για τις τρεις αυτές εκθέσεις. Υπενθυμίζω λοιπόν το χρονοδιάγραμμα. Η προθεσμία για τις τροπολογίες 19 Ιουλίου. Η ψηφοφορία της νομοδότησης της Επιτροπής μας θα γίνει στις 6 Σεπτεμβρίου και η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ θέλει να ψηφίσει τον Νοέμβριο. Θέλει. Έχουμε το σημείο 12 και 13 του κυρίου Γκοντμάνης, αλλά ο κύριος Γκοντμάνης δεν είναι εδώ, αλλά δεν μπορούμε. Έτσι λοιπόν δεν μπορούμε να τις διεκπαιρεώσουμε αυτές τις εκθέσεις σε αναπουσία του. Και ούτως ή άλλως και όλα τα άτομα από την ομάδα του έχουν εξαφανιστεί. Προτείνω λοιπόν να δώσουμε το λόγο στον Γκόραν ε, Φέρμ, ο οποίος είναι ο πιο σοβαρός εδώ πέρα α, βουλευτής που θα κάτσει μέχρι το τέλος και θα σβήσει και τα φώτα. Συνδέονται στην Ευρώπη. Η ομάδα μου είναι... Ναι. μικρή, είπε, δεν έχει εξαφανιστεί τελείως. Ελπίζω, κοιτάξτε, δεν σκοπεύω να κάνω καμία μεγάλη παρουσίαση του μέσου αυτού, γιατί φαντάζομαι πως όλοι γνωρίζετε τι σημαίνει. Απλά να αναφέρω πως, όπως ξέρετε, είναι το νέο ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των διευρωπαϊκών δικτύων μεταφοράς ενέργειας και πληροφορικής. 50 δισεκατομμύρια ευρώ είναι τεράστια αύξηση σε σύγκριση με αυτά τα οποία είχαμε τώρα από αυτά 10 είναι από το Ταμείο Συνοχής, αλλά βεβαίως θα πάνε, είναι δεσμευμένα για τις χώρες συνοχής. Ε, έχω καταθέσει και σκοπεύω να καταθέσω τροπολογίες στη γνωμοδότηση αυτή. Θα σας παρουσιάσω σύντομα το ποιε είναι πρώτα απ' όλα. Είναι οι γνωστές ε, που έχουμε σε όλες αυτές τις γνωμοδοτήσεις. Δεύτερον, προσπαθήσαμε να δούμε το μεγάλο ζήτημα της ανάγκης επενδύσεων που είναι εξαιρετικά σημαντικό. Γι' αυτό είναι προβληματικό γιατί διαβάσαμε κάποια σχόλια ε, επί Προεδρίας Δανίας για το μέσο συνδέοντας στην Ευρώπη ε, που λένε πως εντάξει σημαντικό είναι αυτό αλλά δεν υπάρχει καμία περίπτωση στην κατάσταση που είμαστε τώρα να ακολουθηθούν οι προτάσεις της Κομισιόν. Και το πρόβλημα νομίζω είναι πως ναι, είναι ευκολότερο να γίνουν περικοπές σε νέα μέσα όπου έχουμε νέε φιλοδοξίε από το να κόψουμε μέσα που έχουν ήδη διατεθεί. Είναι ευκολότερο να κόψουμε κάτι το νέο από το να μειωθεί η κοινή γεωργική πολιτική, η πολιτική συνοχή. γιατί αυτά είναι λεφτά που τα έχουν σίγουρα τα κράτη-μέλη ενώ το μέσο αυτό είναι νέες φιλοδοξίες και είναι σημαντικό να μπορέσουμε να αποδείξουμε πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε σε αυτές τις φιλοδοξίες με τους ανάλογους πόρους. Και βεβαίως πρέπει να δούμε και την οξία οικονομική κρίση αλλά και το ότι δεν, υπάρχει, δεν υπάρχουν επαρκείς επενδύσει στην ευρωπαϊκή οικονομία για χρόνια και χρόνια πριν από την κρίση και κάτι πρέπει να γίνει γι' αυτό. Ιδιαίτερα εάν είναι να δημιουργήσουμε μια πραγματική ενιαία αγορά, όχι μόνο από αλλά πραγματική ολοκλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Τότε απαιτούνται αυτές οι επενδύσεις και, να, και σκοπεύουμε να το τονίσουμε αυτό. Το πιο τίμαχο θέμα ήταν τα 10 δις του Ταμείου Συνοχής για τις χώρες αυτές, γιατί κάποιες ε, χώρες ε, θεωρούν πως μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν για άλλους ε, στόχους όπου δεν έχουν τα ίδια λεφτά. Βεβαίως ε, δεν θα αναφερθώ τώρα στις ε, προθέσεις της Κομισιόν γιατί όλοι είμαστε υπέρ έργων με μια ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία όμως θα έλεγα να δώσουμε κάποια μεγαλύτερη έμφαση στη γεωγραφική ισορροπία όταν μιλάμε στην κατανομή πόρων και βεβαίω είναι σαφές πως κάποιες από τις χώρες αυτές θα χρειαστούν στήριξη από την Κομισιόν ε, και για τα 17 αλλά και να ζητήσουν χρηματοδότηση από το άλλο μέρος του μέσου συνδέοντας την Ευρώπη, γιατί είναι επιλέξιμες και γι' αυτό. Και όπως ε, ακούστηκε σε ένα σχόλιο πριν, για το, τα δημοσιονομικά μέσα. Ε, εντάξει, αυτό βεβαίως αφορά τα πιο ανεπτυγμένα κράτη-μέλη, πιο ανεπτυγμένες χρηματαγορές, αλλά θα είναι δύσκολο ε, για τις ε, άλλες χώρες να αντλήσουν χρήματα από εκεί. Θα προσπαθήσω να αναφερθώ και σε αυτό στην έκθεση γιατί αναγνωρίζω αυτό το κίνδυνο αλλά Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος για τη γεωγραφική ισορροπία και για τις περιπτώσεις αυτές βεβαίως. Τα μέσα αυτά, τα χρηματοοικονομικά, είναι γενικά ένα μέσο που θα καταθέσουμε τροπολογίες γιατί θεωρούν πως είναι εξαιρετικά σημαντικό να βρεθούν λύσεις. Είχαμε τα ομόλογα έργων και τη σχετική έκθεση. και κάποια κομμάτια μπήκαν εδώ πέρα στην έκθεση συνδέοντας την Ευρώπη. Θα δούμε επίσης το πώς θα αναμειγνύουμε διάφορα μέσα και διάφορων, ε, διαφόρων ειδών ε, τέτοια μέσα. Και βέβαια πρέπει να κοιτάμε το μέλλον ε, όπως ακριβώς αναφέρεται και στην έκθεση να ανοίγουμε τουλάχιστον την πόρτα σε πιο φιλόδοξα οικονομικά μέσα, όπως παραδείγματο χάρη τα ομόλογα έργων που είναι σε μια πιλωτική φάση ακόμα. Θα προσπαθήσουμε να το αναπτύξουμε λίγο παραπάνω στην έκθεση. Επίσης υπάρχουν κάποιες πιο τεχνικές πτυχές, ε, θα προσπαθήσουμε να αναπτύξουμε την ιδέα των χαρτοφυλακίων έργου. Η Κομισιόν πρότεινε να είναι δυνατόν να μεταφερθούν κονδύλια από ένα μέρος του μέσου σε άλλο. Βεβαίως, εάν θεωρούν πως οι ανάγκες αυξάνονται στην ενέργεια, αλλά δεν υπάρχει τέτοια ανάγκη στην τομέα των μεταφορών ή τον ε, τομέα των ψηφιακών, ναι, να μπορούμε να κάνουμε προσαρμογές. Αλλά είναι πολιτικό ζήτημα και πρέπει να το κρίνουν οι αρχές του προπολογισμού. Ε, αλλιώς φοβούμε πως θα υπάρχει μεγάλη κριτική κατά της διαδικασίας αυτής. Επίσης θεωρώ πως θα πρέπει να δούμε το πεδίο εφαρμογής μέχρι στιγμής αφορά τις υποδομές αλλά υπάρχουν τομεί τομείς όπου θεωρώ πως μπορεί να διευρυνθεί το πεδίο εφαρμογής παραδείγματος χάρη επενδύσεις σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Εν ολίγης, αυτές είναι οι τροπολογίες που έχουν εισαχθεί εδώ πέρα και βεβαίως ε, αναμένω τα σχόλιά σας και τις λοιπές προτάσεις σας. Ευχαριστώ Γέρον. Υπάρχουν σχόλια ή ερωτήσεις προς την εισηγητή. Σας ε, θυμίζω ότι έχουμε μία προθεσμία λίγο μεγαλύτερη, 3 Σεπτεμβρίου προβλέψαμε να εγκρίνουμε την έκθεση στις 20 Σεπτεμβρίου τον Νοέμβριο στα πλαίσια της Ήτρε. Τελειώσαμε την ημερήσια διάταξη αγαπητοί συνάδελφοι, την εξαντλήσαμε. Ραντεβού στις 6 Σεπτεμβρίου θα έχουμε καμιά δεκαριά ψηφοφορίες. Καλές διακοπές. Ευχαριστώ τους συνεργάτες μας και τους εκπροσώπους ε, των άλλων ε, ε, θεσμικών οργάνων, τους υπαλλήλους του Κοινοβουλίου, τους διερμηνείς φυσικά. Όλοι μας αξίζουμε πια καλές διακοπές ώστε να είμαστε σε φόρμα για το δεύτερο εξάμεινο το οποίο θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλό καλοκαίρι.